Ladies and gentlemen, please Κυρίες και κύριοι, παρακαλώ καθίστε. Καλημέρα σας. Παρά το κυκλοφορικό και τις δυσκολίες πρόσβασης στο Κοινοβούλιο, καλωσορίζω ε, όλους αυτήν την δεύτερη ημέρα της ε, συνεδρίας της Επιτροπής για την Ασφάλεια και την Άμυνα. Έχουμε και άλλα πολύ ενδιαφέροντα σημεία στην ημερήσια διαταξή μα και γι' αυτό θα σα παρουσιάσω αμέσω το πρώτο. Ένα εργαστήριο το οποίο συνήθω έχει ετοιμάσει η Υπηρεσία Πολιτικού Σχεδιασμού με τη βοήθεια της Γραμματείας της Επιτροπής Ασφάλειας και Άμυνας λάβαμε υπόψη πολλά οργανωτικά θέματα που έπρεπε να έχουν λυθεί προηγουμένως και το θέμα είναι οι σχέσεις μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ε, οι σχέσει των Ευρωπαϊκών Κρατών Μελών με τη Σαουδική Αραβία στον τομέα τη ασφάλεια και τη άμυνα. Θα ήθελα να σα παρουσιάσω τι δύο προσκεκλημένε μα, την κυρία Νιέ Λεβαλουά, η οποία είναι ε, ερευνήτρια και καθηγήτρια. σε ίδρυμα που έχει την έδρα του στο Παρίσι για στρατηγικές έρευνες και δεύτερος, δεύτερη μάλλον, η κυρία Τζέιν Κίνεμαντ, η οποία είναι ερευνήτρια επίσης σε ένα γνωστό think tank η οποία ασχολείται με τα προβλήματα της Μέσης Ανατολής και της ε, Βόρειας Αφρικής. Καθώς έχουμε καθυστερήσει λίγο, και φαντάζομαι ότι θα κατακλείσουν την αίθουσα οι θεατές να, εντός ολίγου να ξεκινήσουμε αμέσως. Πρώτα απ' όλα να δώσω το λόγο στην καθηγήτρια Νιές Λεβαλουά και μετά στην κυρία Τζέιν Κινέμαντ. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Μιλήσαμε σήμερα το πρωί, αναφέρατε μάλλον, θα μιλήσουμε για την Σαουδική Αραβία και τις ανάγκες της σε άμυνα και ασφάλεια στο βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας και να δούμε γιατί το βασίλειο αυτό έχει ανάγκη από ασφάλεια και από άμυνα. Νομίζω το πρώτο που πρέπει να κοιτάξουμε είναι γιατί υπάρχει αυτή η σοβαρή ανάγκη ασφάλειας και άμυνας, ποιοι είναι οι λόγοι που προξενούν αυτή την ανάγκη και ο πρώτος λόγος είναι να λάβουμε υπόψη το ευάλωτο του, σαουδικού, του καθεστώτος. Η Σαουδική Αραβία είναι ένα βασίλειο που προφανώς αισθάνεται ευάλωτο, έχει τροτά σημεία και γι' αυτό χρειάζεται να επενδύσει μαζικά στην ασφάλεια για να εξασφαλίσει, θα έλεγα, μια ασφάλιση, να αγοράσει τρόπο την μια ασφάλεια ζωή και να επιβιώσει σε ένα εχθρικό περιβάλλον και να αισθανθεί ε, ανακούφιση. Γιατί μιλάμε για ευάλωτο στην περίπτωση του βασιλείου τη Σαουδική Αραβία. Πρώτα απ' όλα, νομίζω, λόγω των συνθήκων ε, εντό των οποίων γεννήθηκε το βασίλειο αυτό. Ε, την συμφωνία μεταξύ μιας οικογένειας, της οικογένειας Σαούντ και των θρησκευτικών ε, υπόλοιπων ομάδων, οι οποίοι δημιούργησαν ένα σύμφωνο για τη δημιουργία αυτού του βασιλείου. Η οικογένεια Σαούντ και οι διάφορες θρησκευτικές ομάδες και οι οποίες ε, έχουν να κάνουν με το πώς η βασιλική οικογένεια δέχεται τη θρησκευτική διοργάνωση της χώρας, η οποία βέβαια θρησκευτική δομή δεν έχει αναγκαστικά την ίδια άποψη για το πώς θα πρέπει να εξελιχθεί η χώρα, όπως η βασιλική οικογένεια. Το δεύτερο είναι οι γειτονικέ χώρες στη γεωγραφική αυτή περιοχή. Η Σαουδική Αραβία βρίσκεται σε ένα περιβάλλον ιδιαίτερα ε, ταραγμένο, με, την, με τον πόλεμο στην Ιεμένη, θα το ξαναδούμε, αλλά και με τα εσωτερικά προβλήματα. Ξέρετε ότι η Αραβία έχει δεχτεί πολλές επιθέσεις, σοβαρές επιθέσεις, Πράγμα που δείχνει τις δυσκολίες αυτού του βασιλείου. Βεβαίω, την επαύριο ε, κάποιων επιθέσεων, ε, το βασίλειο αυτό έλαβε ισχυρά μέτρα ο κληρονόμος πρίγκιπας ε, ανέλαβε το θέμα βέβαια αυτό και έδειξε ότι τα τελευταία χρόνια έχει τη δυνατότητα να αντιμετωπίσει τις εσωτερικές πιέσεις που παρουσιάζονται από τις θερμοκρατικέ επιθέσεις κατά της Σαουδικής Αραβίας σήμερα και του Ισλαμικού κράτους που αυτή τη στιγμή έχει παρουσία στο Βασίλειο παρόλο που ακόμα δεν έχει αναλάβει δράση. Είναι όμως μια οργάνωση που σήμερα στοχεύει και τη βασιλική οικογένεια θεωρώντας ότι δεν σέβεται τις ε, βασικές αξίες του Ισλάμ και δεν μπορεί να παρουσιάζεται ως ο εκπρόσωπος, ο επίσημος εκπρόσωπος του Ισλάμ. Ξέρετε ότι ε, βρίσκονται οι ιερές πόλεις του Ισλάμ στη Σαουδική Αραβία, η Μέγα και η Μεδίνα, ή έχουν πολλά παρακλάδια στην περιοχή αυτή η Αλκάιντα της Σαουδικής Αραβίας και το τμήμα του Ισλαμικού κράτους που δραστηριοποιείται εκεί. Η συμφωνία λοιπόν που έχει επιτύχει η Σαουδική Αραβία για τη δημιουργία της αλλά και οι συμφωνίες που έχει με το Ιράν είναι πολύ ε, η Σαουδική Αραβία ανισχύει για την ενδεχόμενη επιστροφή του Ιράν στο διεθνέ προσκήνιο. Είναι μια μεγάλη δύναμη τη περιοχή που θα μπορούσε να δυσκολέψει την περιφερειακή αυτή δύναμη που εκπροσωπεί η ίδια η Σαουδική Αραβία. Η συμφωνία μεταξύ του λοιπόν για την Αραβία θεωρείται ω μια πρόκληση. Μια πρόκληση την οποία πρέπει να αντιμετωπίσει εφόσον το Ιράν επιστρέψει στην, στο διεθνές προσκήνιο ιδίω με τα ζητήματα του πετρελαίου που τίθενται, διότι από το εμπάργκο και μετά ε, η παραγωγή του Ιράκ περιορίστηκε πάρα πολύ, έτσι η Σαουδική Αραβία μπόρεσε να καθορίζει την διεθνή αγορά πετρελαίου, να έχει μια ισχυρή θέση εκεί, ανάλογα με τα συμφέροντά τη. Με την άφηξη βεβαίω του Ιράν τα πράγματα αλλάζουν και πέραν του πώ θα διαχειρίζεται την αγορά του πετρελαίου, ένα άλλο ερώτημα που τίθεται για τη Σαουδική Αραβία είναι το κατά πόσο μπορεί να αντιμετωπίσει απέναντί τη ένα κράτο που θα αρχίσει να επενδύει, να έχει περιφερειακέ φιλοδοξίε, περι... φιλοδοξίε δηλαδή στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή. Το Ιράν που θα διεκδικήσει τη θεμητή του, όπω θεωρεί θέση στην όλη γεωγραφική περιοχή και στο διεθνέ προσκήνιο. Η συμφωνία λοιπόν αυτή δημιουργεί ένα μείζον πρόβλημα για του Σαουδάραβε, διότι θεωρούν ότι η συμφωνία με το Ιράν μπορεί να θέτει ένα αμφιβόλο την ε, αδιάρρηκτη, σχέση που έχει το, το Ριάντ με την Ουάσιγκτον. Ε, Είναι σημαντικό λοιπόν αυτό για το βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας που αισθάνεται εν μέρη ότι τον εγκαταλείπει ε, ο Αμερικανός σύμμαχός του. Οι Σαουδάραβες πραγματικά ξαφνιάστηκαν από τον τρόπο με τον οποίο οι Αμερικανοί παράτησαν τους άλλους συμμάχους τους στην περιοχή. Όπως ε, τον κύριο Χαλίλ τον Ίσιο ή τον κύριο Μουμπάρακ, τον Αιγύπτιο. Οι Σαουδάραβε δεν φαντάζονταν ότι θα παρατούσαν τόσο εύκολα τον Μουμπάρακ οι Αμερικανοί που ήταν ένα μεγάλο του σύμμαχο, Εάν μπορούν να φέρονται στον Μουμπάρακ με αυτόν τον τρόπο, σκέφτηκαν τη μέρα που ο θρόνο θα διεκδικηθεί από άλλε δυνάμει ή θα υπάρξει κάποια ταραχή στη χώρα, φανταστείτε τι θα γίνει. Τώρα οι Σαουδάραβε έτσι βλέπουν και την συμμαχία του με του Αμερικανού συμμαχία που ξεκίνησε στη δεκαετία πριν αρχίσουν οι αμφισβητήσεις και οι εξεγέρσεις στον αραβικό κόσμο. Όλα αυτά λοιπόν έχουν να κάνουν με το πώς αντιλαμβάνεται η Σαουδική Αραβία τις ε, δικές της αδυναμίες και για την έφραυστη εσωτερική πολιτική κατάσταση πρέπει να μιλήσω. Έχει και αυτή σχέση με το πώς αισθάνεται ευάλωτη η Σαουδική Αραβία. Μιλάμε για την αντιπαλότητα που χωρίζει τον ε, τον ε, κληρονόμο πρίγκιπα και τον ε, τον Μοχάμεντα Γεφ ο οποίος έχει ασχοληθεί με την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και ο οποίος έχει μια ιδιαίτερη φήμη, χέρι εκτίμησης από τους Σαουδάραβες, διότι έχει νομιμοποίηση στο, στη θέση που καταλαμβάνει, ενώ ο αντίπαλός του που είναι μόλις 35 ετών και ο οποίο έχει αναλάβει το χαρτοφυλάκιο τη άμυνα, ένα πολύ σημαντικό υπουργείο για τη χώρα, έχει έρθει και αυτό με τις φιλοδοξίες του και πρέπει και αυτό να αποδείξει ότι αξίζει τη θέση του στη βασιλική οικογένεια, στη Σαουδική Αραβία, να δείξει ότι νομιμοποιείται στη θέση που καταλαμβάνει ω υπουργό άμυνα. Δηλαδή είναι Είναι και αυτός κληρονόμος στο βασιλικό θρόνο και έχει αυτήν την ε, ιδιαίτερη θέση του Υπουργού Άμυνας. Πρέπει λοιπόν έτσι να εκτιμήσουμε την εμπλοκή της Σαουδικής Αραβίας στον πόλεμο της Ιεμένης. Ο Μοχάμεντ Μπεν Σαλμάν, ο υπουργό τη Άμυνα, είναι ένα άνθρωπο αρκετά ισχυρό. Ο πόλεμο αυτό του δείχνει την ευκαιρία να επιβεβαιώσει τη θέση του υπουργού Άμυνα και να δείξει ότι έχει την πυγμή για να διεξάγει τι επιχειρήσει στην Ιεμένη και να λάβει αυτή την νομιμοποίηση που αυτή τη στιγμή δεν έχει, την αναγνώριση που, που θεωρεί ότι του χρειάζεται. Ο πόλεμος λοιπόν στην Ιεμένη θα βελτιώσει τη θέση του και στο επίπεδο της βασιλικής οικογένειας και μεταξύ των Σαουδαράβων. Η εμπλοκή τη Σαουδική Αραβία ξεκίνησε το Μάρτιο του 2015, ένα μισή χρόνο τώρα. Για την ώρα δεν βλέπουμε να έχει επιτευχθεί κανένα αποτέλεσμα. σα ίσα που ο πόλεμο μένεται. Οι πρωτοβουλίε για ειρήνη, οι διαπραγματεύσει που κατέληξαν έτσι καλώ σε αδιέξοδο τον περασμένο Αύγουστο δεν οδήγησαν σε αποτέλεσμα και βλέπουμε να συνεχίζεται το εμπάργκο και η κατάσταση στην Εμένη να γίνεται ολοένα και χειρότερη και ολοένα και πιο δραματική για τον τόπιο πληθυσμό. Μάλιστα, στο έδαφο τη Ιεμένης δραστηριοποιούνται πλέον ριζοσπαστικέ ομάδε που υποφελούνται από τις ε, συνθήκε πολέμου, ιδίω από την Αλκάιντα τη Σαουδική ε, Χερσονήσου, Χερσονήσου και το ΝΤΑΕΣ, το που στο παρακλάδι του στη Σαουδική Σαουδαραβική Χερσόνησο, κοιτάζει να παρισφρήσει από εκεί για να περάσει μετά στη Σαουδική Αραβία. Βλέπουμε τώρα τις αδυναμίες της Σαουδικής Αραβίας, καταλαβαίνουμε γιατί η Αραβία έχει αυτήν την τόσο σημαντική ανάγκη εξοπλισμού και αγοράς αμυντικού εξοπλισμού ανά τον κόσμο. Θέλει να δημιουργήσει ένα προστατευτικό, ε, ε, μια προστατευτική ασπίδα γύρω της, για να προστατευθεί από τις εσωτερικές της αδυναμίες, τις αδυναμίες της στην δική της γεωγραφική περιοχή και το διεθνές προσκήνιο. Έτσι αισθάνονται οι Σαουδάραβες σήμερα απέναντι στους Αμερικανούς. Δεν θέλω να πω βέβαια ότι οι Αμερικανοί θα πετάξουν από τη μια στιγμή στην άλλη, στην άκρη, το βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας. Τους χρειάζονται και θέλουν να είναι σταθεροί οι Αμερικανοί είναι ένα σημαντικό σύμμαχο και δεν σημαίνει ότι επειδή οι Αμερικανοί ανέλαβαν πρωτοβουλία στην υπογραφή τη συμφωνία με το Ιράν θα παρατήσουν του Σαουδάραβε. Όμω αυτή η ανασφάλεια των Σαουδαράβων πρέπει να ληφθεί υπόψη για να καταλάβουμε πώς σήμερα η Σαουδική Αραβία προσπαθεί απεγνωσμένα να αγοράζει όπλα ανά τον κόσμο για να εξασφαλίσει την ασφάλειά τη. Αυτό που πρέπει να καταλάβουμε βέβαια είναι ότι η Σαουδική Αραβία σήμερα, και αυτό είναι ένα άλλο στοιχείο που επιτρέπει να καταλάβουμε τη στρατηγική της και ακριβώς την αγορά αμυντικού εξοπλισμού και τη διόγκωση του στρατιωτικού υλικού που διαθέτει, είναι ότι σήμερα η Σαουδική Αραβία έχει έρθει στο προσκήνιο τη δική τη γεωγραφική περιοχή ω η μόνη δύναμη που μπορεί να αναλάβει δράση τα προηγούμενα χρόνια. Κυρίω πριν την έναρξη των Αραβικών Επαναστάσεων, ήταν σαφέ ότι οι περιφερειακέ δυνάμει ήταν η Αίγυπτο, οι ισχυρέ δυνάμει, ήταν η Αίγυπτο, παρόλο που τα τελευταία χρόνια ο Χωσέ και είχε χάσει λίγο το κύρο του και τη δυνατότητα να μπορεί να είναι παρόν οπουδήποτε, στο περιφερειακό προσκήνιο. Όμω η Αίγυπτο είχε το φυσικό ρόλο τη περιφερειακή δύναμη στη Μέση Ανατολή με τη δυνατότητα να μπορεί να παίρνει θέση, να διαμεσολαβεί, να διαχειρίζεται την κατάσταση της ευρύτερης περιοχής. Με την Επανάσταση όμως ε, στην Αίγυπτο, με την ε, άφηξη του Μόση, με τις υπόλοιπες εξελίξεις στην Αίγυπτο, η Αίγυπτος έχει πρώτα απ' όλα εσωτερικά προβλήματα. Δεν έχει την ε, το χρόνο και την ε, διαθεσιμότητα να ασχοληθεί με τα προβλήματα της ευρύτερης περιοχής. Στη Συρία ξέρετε τι γίνεται σήμερα. Είναι στο, σε χάος και σε πόλεμο. Το Ιράκ μετά την Αμερικανική εισβολή επίσης βρίσκεται σε απόλυτο χάος. Εάν δούμε λοιπόν την ευρύτερη γεωγραφική περιοχή, ποια είναι η μόνη περιφερειακή δύναμη που μπορεί να αναλάβει αυτό το ρόλο, είναι η Σαουδική Αραβία. Είναι η μόνη χώρα που σήμερα μπορεί να αναλάβει κάποιο ρόλο η Αραβία όμω δεν θέλει να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο. Ήθελε να είναι δευτεραγωνίστρια και να έχει έμεση εμπλοκή σε όλα τα θέματα. Τώρα ξαφνικά έχει σπροχτεί μπροστά στη σκηνή και πρέπει να παίξει το ρόλο τη ω περιφερειακή δύναμη. Βλέπουμε λοιπόν να δραστηριοποιείται σε διάφορε περιοχέ στη Συρία όπου είχε ένα σημαντικό ρόλο ή τουλάχιστον θέλησε να παίξει ένα σημαντικό ρόλο υποστηρίζοντα τι θέσει που ξέρουμε. Αυτή τη στιγμή η σαουδική πολιτική προς τη Συρία έχει δημιουργήσει προβλήματα. Μετά την ρωσική εισβολή του Ιράν και της, της Χεσμολάκ, βλέπουμε τι συμβαίνει, βλέπουμε τη σχέση της με το καθεστώς του, του και την ε, δική της ε, τοποθέτηση. Η Σαουδική λοιπόν Αραβία ξαφνικά βρίσκεται να έχει εμπλοκή στις περιφερειακές ε, συγκρούσεις και δυσκολεύεται να έχει μια πραγματική πολιτική θεώρηση των πραγμάτων, ένα πολιτικό όραμα, ώστε αυτό το όραμα να λειτουργήσει και στην πραγματικότητα και να της επιτρέψει να παίξει αυτό το ρόλο. Τι συμβαίνει λοιπόν σήμερα. Έχουμε μια Σαουδική Αραβία με πολλές αδυναμίες, όπως σας την παρουσίασα. Επίσης πρέπει να δραστηριοποιηθεί ως σου παράγοντας. Επίσης είναι εμπλεγμένη στην περίπτωση της Ιεμένης με τα αποτελέσματα που βλέπουμε με πολλά προβλήματα χωρίς να υπάρχουν αποτελέσματα. Η Σαουδική Αραβία λοιπόν φτάνει να πει τι κάνω τώρα, πώς να ε, πράξω. Η Σαουδική λοιπόν Αραβία προσπαθεί να διαφοροποιήσει τις πηγές από τις οποίες αντλεί αμυντικό εξοπλισμό. Περνάει σε συμφωνίε με άλλες χώρες πέρα από το φυσικό τη σύμμαχο που είναι οι ΗΠΑ, με, με τι οποίε υπάρχει μια καχυποψία στις σχέσεις ανοίγει τη Σαουδική Αραβία, διαφοροποιεί τις πηγές της. προς την ε, Ρωσία κυρίως με την επίσκεψη του Πούτιν ε, στην, ε, στο Ριάντ που ήταν κάτι το πρωτοφανές αλλά και με τους Ευρωπαίους οι οποίοι θέλουν να ενισχύσουν την προσπάθεια των Σαουδαράβων να διαφοροποιηθούν η Γαλλία εδώ και χρόνια έχει μια πολύ σοβαρή πολιτική κίνηση προς τη Σαουδική Αραβία, προσπαθώντας να επαναθερμάνει τις σχέσεις με αμυντικές συμβάσεις που έχουν ήδη υπογραφεί. Τώρα πρέπει να δούμε βέβαια μεταξύ της ε, αναγγελίας αμυντικών ε, συμβάσεων και αγορών κατά πόσον θα πραγματοποιηθούν αυτές. Υπάρχει πάντα μια απόσταση μεταξύ των δύο. Όμω, αυτή τη στιγμή υπάρχει βούληση από κάποιε ευρωπαϊκέ χώρε, από την Γαλλία, τη Μεγάλη Βρετανία, τη Γερμανία, που αρχίζει να μπαίνει στο παιχνίδι, γιατί πολλά χρόνια τώρα η Γερμανία ήταν πολύ επιφυλακτική. Δεν ήθελε να παραδίδει εξοπλισμό σε χώρε οι οποίε μπορεί να είχαν κρίση, προβλήματα. Σήμερα όμω βλέπουμε ότι η Γερμανία να αρχίζει να ενδιαφέρεται για την αγορά τη Σαουδική Αραβία. Για λόγου προφανεί βεβαίω, διότι η Σαουδική Αραβία έχει χρήμα. Και θέλει να αγοράσει αμυντικό εξοπλισμό. Το ερώτημα λοιπόν που τίθεται σήμερα είναι σε ποιο βαθμό θα καταφέρει η Σαουδική Αραβία να διαφοροποιήσει τι πηγέ ε, ανεφοδιασμού τη. Είδαμε τα τελευταία χρόνια ότι έχει διάθεση να διαφοροποιήσει, να διευρύνει του οριζοντέ τη και το κάνει. Δεν πρέπει όμω να τα πατώμεθα και να πιστεύουμε ότι τα πράγματα θα αλλάξουν ριζικά Υπάρχει αυτή η διάθεση, αυτή η επιθυμία των ε, Σαουδαράβων να δείξουν ότι είναι σχετικά ανεξάρτητοι από του Αμερικανού. Θέλουν να έχουν αμυντικέ σχέσει αγορά εξοπλισμού με άλλε χώρε. Οι Αμερικανοί όμω παραμένουν ο ουσιαστικό κατά προτεραιότητα σύμμαχο τη Σαουδική Αραβία, διότι το μεγαλύτερο μέρο των εξοπλισμών προέρχονται από τι ε, ΗΠΑ και βεβαίω η στρατιωτική τη Σαουδική Αραβία κυρίω εκπαιδεύοντα τι ΗΠΑ. Δεν αλλάζει από την μέρα στην άλλη δηλαδή ο φυσικό σύμμαχο μια τέτοια χώρα, στον τομέα τη άμυνα ιδίω. Είναι πολύ σοβαρέ οι υποδομέ που έχουν γίνει σχετικά και οι προβλέψει. Δεν αλλάζουν αυτά από την μέρα στην άλλη. Δηλαδή οι Σαουδάραβε λένε του Αμερικανού, κοιτάξτε, ακόμη και αν έχουμε πολύ στενέ σχέσει, μπορούμε να κάνουμε και άλλα πράγματα και κάπω προσπαθούν να αυτονομήσουν την αμυντική του πολιτική. Όμω, παρόλα αυτά, αυτέ οι προσπάθειε αυτονόμηση είναι πολύ περιορισμένε. Δηλαδή δεν μπορεί να γίνει τώρα στροφή 180 μοιρών. Θα χρειαστεί χρόνο. Το τελευταίο σημείο που ήθελα να θίξω και μου φαίνεται ενδιαφέρον είναι πώ αντιδράει η κοινωνία τη Σαουδική Αραβία όλα αυτά. Νομίζω η τάση, όταν μιλάμε για τι χώρε τη Αγγλία και Μέση Ανατολή, είναι να μιλάμε για κράτη, συγκρούσει, εντάσει, το χάο που επικρατεί. Είναι μια πραγματικότητα αυτό, αλλά υπάρχουν και κοινωνίε που ζουν σε αυτά τα κράτη. Πρέπει λοιπόν να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε πώ οι Σαουδάραβε αντιδρούν και αντιλαμβάνονται όλη αυτή την κατάσταση. Οι Σαουδάραβε, τουλάχιστον ένα μέρο αυτών, διαρωτώνται σε τι ε, χρησιμεύουν όλα αυτά τα μυθόδη ποσά που ε, εκταμιεύει η βασιλική οικογένεια για να προστατευτεί, με αποτελέσματα που δεν φαίνεται να είναι και πολύ αυτά. Δηλαδή, θυμηθείτε, όταν έγινε ο πόλεμο στο Ιράκ, παρόλο που οι Σαουδάραβε είχαν επενδύσει εκατοντάδε ε, δι δολάρια στον εκπλησμό του, ζήτησαν εξωτερική βοήθεια για να προστατευτούν τοπικό λοιπόν πληθυσμό αναρωτιέται γιατί αυτέ οι δαπάνε, αφού ούτω ή άλλω η Σαουδική Αραβία αισθάνεται πάντοτε και ακόμα ευάλωτη. Και διαρκώ ε, παρεκτρέπεται, διαρκώ μάλλον εκτροχιάζει την ε, βασική τη πορεία ανεξαρτησίας προ την έκκληση βοήθεια στου εξωτερικού συμμάχου. Αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη, διότι οι δράσει τη ε, τοπική κοινωνία τη Σαουδική Αραβία μπορεί να επηρεάσει τα πράγματα, γιατί διαρκώ εντείνεται. Οι Σαουδάραβες πολίτες ε, γνωρίζουν αυτή τη στιγμή τι συμβαίνει, ενημερώνονται, μπορεί να αντιδράσουν και μπορεί και να εγκαλέσουν τους εθνοντέ του για την ε, διαχείριση των πόρων της χώρας. Και αυτό ακόμη περισσότερο διότι λόγω της πτώσης των τιμών του πετρελαίου η αναδιανομή που είναι πολύ σημαντικότερη από τα προηγούμενα χρόνια και με το σύμφωνο που υπάρχει μεταξύ βασιλικής οικογένειας και σαουδικής ε, κοινωνίας το οποίο είναι εμείς θα σας κυβερνάμε να σας δώσουμε τα μέσα για να ζείτε καλά, έχουμε το χρήμα του πετρελαίου και θα το μοιράζουμε σωστά. Εάν λοιπόν αυτό το χρήμα είναι λιγότερο διαθέσιμο γιατί υπάρχει λιγότερο χρήμα, πέφτουν οι τιμές του πετρελαίου και ο πληθυσμός αυξάνεται ταυτόχρονα, η αναδιανομή αυτών των πόρων, των κερδών θα περιοριστεί. Εκεί μπορεί να αρχίσει να εκφράζει διεκδικήσει και αιτήματα η κοινωνία τη Σαουδική Αραβία. Αφού το αρχικό σύμφωνο τίθεται να αμφιβόλα, αφού έχουμε λιγότερο χρήματα, εποφελούμαστε λιγότερο από την αναδιανομή του πλούτου του πετρελαίου, μπορεί και να θελήσουμε να έχουμε πρόσβαση στην πολιτική, να, εκφράσουμε, να εκφράσουμε κάποιες πολιτικές διεκδικήσεις. Αυτό είναι ένα στοιχείο που μακροπρόθεσμα μπορεί να αποσταθεροποιήσει το πολιτικό σύστημα όπως έχει διαμορφωθεί. Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να δείξουμε ιδιαίτερη προσοχή σήμερα σε αυτά που εκφράζει η κοινωνία τη Σαουδική Αραβία για το πώς διαχειρίζεται του πόρου της χώρας η βασιλική οικογένεια, ιδίω για την άμυνα ε, και την ασφάλεια που ε, ε, αφομοιώνει και απορροφά τεράστια ποσά από τον προπολογισμό της χώρας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η παρουσίαση και τώρα θα δώσω το λόγο στην κυρία Τζέιν Κίνινμοντ από το Chatham House. Ευχαριστώ πολύ. Σήμερα η Σαουδική Αραβία είναι η δεύτερη μεγαλύτερη αγορά εξαγωγών όπλων από την Ευρωπαϊκή Ένωση μια ευρωπαϊκή χώρα μετά από τη ΣΥΠΑ και έχει υπάρξει, αν θέλετε, μια δραματική εμβάθυνση και επέκταση των σχέσεων άμυνα και ασφάλεια μεταξύ Σαουδική Αραβίας και βασικών ευρωπαϊκών κρατών τα τελευταία 15 χρόνια. Ήδη, μάλλον ακόμη η περιορισμένη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση και το περιφερειακό μπλοκ, ε, το Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπη, παραμένει αλλά η σχέση μεταξύ ε, των δύο αυτών οργανώσεων εστιάζει στις εμπορικές σχέσεις. Βέβαια, έχει συζητηθεί για δύο δεκαετίες το θέμα μια συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών χωρίς να προχωρήσει. Αλλά στο περιφερειακό επίπεδο λίγη είναι η εστίαση στη συνεργασία σε θέματα άμυνας και ασφάλειας και υπάρχει μια μεγάλη αντίθεση μεταξύ αυτών τη της περιφερειακής θεσμικής συνεργασίας και των δημερών σχέσεων μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και με μονομένα κρατομέλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου τα ευρωπαϊκά κράτη-μέλη ουσιαστικά ανταγωνίζονται μεταξύ τους σε μεγάλο βαθμό για το να είναι σύμμαχοι, εταίροι και πάροχοι όπλων και άλλων εξοπλισμών στη Σαουδική Αραβία πολύ δύσκολα συνεργάζονται μεταξύ τους για να μεγιστοποιήσουν τα κοινά ευρωπαϊκά συμφέροντα όπως αναπτύσσονται οι πολιτικές της Σαουδικής Αραβίας. Μετά το boom στο ντομά του πετρελαίου το 2011, οι αμυντικές δαπάνες ε, της Σαουδικής Αραβίας αυξάνονταν συνεχώς. Είναι Ήταν μια εποχή όμως που συνοδευόταν και με μεγάλη πολιτική αγωνία, όπως είπε και η Ανιές, ιδίως λόγω των ε, αναταχών στο Ιράκ. Και υπάρχει γενικά μια ανησυχία για το ρόλο του Ιράκ. Και είχαμε και την Αραβική Άνοιξη, τις εξεγέρσεις της αραβικές χώρες και τις διάφορες επιπτώσεις που επηρέασαν. Και βέβαια έχουμε και το ISIS είναι απειλή και για τις ευρωπαϊκές χώρες και για τη Σαουδική Αραβία, όπου έχει φέρει σε πέρας σημαντικές βομβιστικές επιθέσεις. Αυτά είναι το υπόβαθρο. Η Σαουδική Αραβία ζητά πιο βαθιές σχέσεις άμυνας και ασφάλειας και πιο ποικίλε σχέσεις, δηλαδή πέραν των παραδοσιακών σχέσεων με ΙΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο και Γαλλία, αναστικά του παραπάνω. Και έτσι έχει αναπτύξει στενότερους δεσμούς με μια σειρά άλλων ευρωπαϊκών κρατών και δυτικών και ανατολικοευρωπαϊκών. Ταυτόχρονα όμως προκύπτουν κάποια ερωτήματα για το βαθμό στον οποίο ευρωπαϊκές χώρες και η Σαουδική Αραβία έχουν κοινά συμφέροντα στη Μέση Ανατολή και κατά να αντιλαμβάνονται με τον ίδιο τρόπο το τι θα πει σταθερότητα και ασφάλεια στην περιοχή αυτή. Αυτές οι διαφορές έχουν έρθει στο προσκήνιο με τον πόλεμο στην Ιεμένη πολύ περισσότερο, πολύ πιο έντονα από ό,τι μέχρι τώρα. Πριν τις εξεγέρσεις ε, στην ε, σε αραβικές χώρες το 2011. Πολλές χώρες θεωρούσαν ότι η Σαουδαραβική κυβέρνηση ήταν μια συντηρητική δύναμη σε ό,τι αφορά να μην και την ασφάλεια, δηλαδή ότι προσπαθούσε πιο πολύ να διατηρήσει την ε, νομιτάξη, αν θέλετε. Και αυτό ευθυγραμμιζόταν σε μεγάλο βαθμό. Με τα βασικά συμφέροντα άμυνας και ασφάλειας της Ευρώπης και των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο αντίκτυπος θρησκευτικών δικτύων της Σαουδική Αραβίας είναι λίγο πιο πολύπλοκο θέμα. Εδώ νομίζω ότι πρέπει να τονίσουμε ότι η κυρίαρχη ερμηνεία του Ισλάμ στη Σαουδική Αραβία είναι επίσης συντηρητική, παραδοσιακή. Ουσιαστικά επιθυμεί μια πολιτική σταθερότητα, ηρεμία. Δεν ερμηνεύει το Ισλάμ ως κάτι το οποίο προωθεί, εγκομιάζει και ορειοποιεί ε, επαναστάσεις. Ωστόσο υπάρχει και ο σαλαφισμός εκεί που αποτέλεσε κάποτε πρόσφαρο έδαφος για ορισμένες φορές επαναστατικές τσιχαντιστικές ομάδες. Υπάρχουν λοιπόν πραγματικά δικαιολογημένες ανησυχίες για το ρόλο των θρησκευτικών δικτύων αυτών ε, σε ό,τι αφορά στην Ευρώπη και αλλού. Και αυτό βέβαια είδαμε να δημιουργεί ιδιαίτερε εντάσει μεταξύ Σαουδική Αραβία και Ηνωμένων Πολιτειών μετά την επίθεση 11 Σεπτεμβρίου και πρόσφατα πάντα ε, στην ε, στις ΗΠΑ σχέση με τον ΤΑΕΣ. Αυτά βέβαια δεν εντάσσονται ε, στο μεγαλύτερο μέρος τους στην αμυντική πολιτική, στην εξωτερική πολιτική. Όμως υπάρχουν άλλοι μη κρατικοί παράγοντες που κινητοποιήθηκαν πολλές φορές, ε, ιδίως στο Αφγανιστάν 1980, μια πολιτική που στηρίχθηκε τότε βέβαια και από τη ΣΥΠΑ και πιο πρόσφατα στη Συρία για στόχους εξωτερικής πολιτικής. Όμως μετά τις εξεγέρσεις ε, του 2011 στις αραβικές χώρες η ε, πολιτική αυτή αναταραχή στη Μέση Ανατολή έχει ενθαρρύνει τη χώρα να ακολουθήσει μια ε, πιο επιθετική προσέγγιση, πιο επαναστατική προσέγγιση στα περιφερειακά, στις περιφερειακές συγκρούσεις. Και αυτό ενισχύθηκε με την όνομα του εξουσία ενός νέου ηγέτη, Σαουδική Αραβία. Όμως αντικατοπτρίζει και το γεγονός ότι δεν είναι δυνατόν η χώρα να παρακολουθεί απλά και να διατηρεί το status quo με ένα συντηρητικό τρόπο. Γιατί δεν υπάρχει και status quo πλέον στην περιοχή. Σε κάποιο βαθμό όλοι έχουν αναγκαστεί να πάρουν ε, μια θέση. Η κατάσταση είναι γενικά ρευστή και εξελίσσεται. Και έχουμε δει και η ευρωπαϊκή πολιτική να αλλάζει συν το χρόνο σε ό,τι αφορά αυτές τις εξεγέρσεις, ιδίω σε σχέση με τη Σύρια. Που είναι πολύ δύσκολο να καταλάβει κανείς τελικά και ποια είναι ε, στη βάση της αυτή η ευρωπαϊκή πολιτική. Η προσέγγιση της Σαουδικής Αραβίας έχει επηρεαστεί και από αυτό που αντιλαμβάνω πολλαπλές απειλές, ε, τα κάλυψε η Ανία σε μεγάλο βαθμό αυτά. Υπάρχουν φόβοι ενός μεγάλου κένου ασφαλείας, τάξης και εξουσίας στην περιοχή. Λόγω του ότι έχουν καταρρεύσει τα παραδοσιακά κέντρα ισχύω και νομίζω ότι όταν προσπαθούμε να καταλάβουμε αυτές τις αντιλήψεις και ιδέες στη Μέση Ανατολή θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι μπορεί να νιώθει και μεγάλη γωνία Ευρώπη για την κρίση, την προσφυγική. Όσοι όμως ζουν ε, στη Μέση Ανατολή, το ζουν από πολύ πιο κοντά όλο αυτό το φαινόμενο. Το ζουν, ε, είναι βιωματικό. Ε, καθότι έχουν καταρρεύσει κράτη και βλέπουν πολύ πιο έντονο αυτό το φαινόμενο. Η Σαουδική Αραβία ταυτόχρονα ανησυχεί για το ότι είπα πια είναι πιο ξεκάθαρη, δεν είναι αμφίσιμη η στάση της ό,τι αφορά και την παρουσία της στη Μέση Ανατολή. Ένα από τα ζητήματα που αφορούν τις μελλοντικές προοπτικές και τα ερωτήματα είναι αυτό το φαινόμενο της κυβέρνησης Ομπάμα μόνο ή όχι. Η ελίτ Ψωτική Αραβία δεν έχουν πολύ ξεκάθαρη άποψη Μπορεί να μην είναι θετικέ οι απόψει αλλά δεν είναι και σαφέ. Αν ο επόμενο πρόεδρο των υπόπτη και αν είναι, ή όποια και αν είναι, θα συνεχίσει τι ίδιε πολιτικέ. Και η Σαουδική Αραβία αγωνιά επίση για το μήπω αυτό το κενό ασφάλεια και ε, εξουσία εν μέρη, μήπω το αντιληφθεί και το εκμεταλλευτεί το Ιράν και γύρω από, αυτή, ε, γύρω από αυτό. Οι αμυντικές δαπάνες σας είπα ότι ήταν αυξημένες τα τελευταία 15 χρόνια και αυτό κυρίως λόγω του φόβου του Ιράν και ίσως είναι ηρωνικό αυτό, αλλά πολλές ευρωπαϊκές χώρες έχουν αποφεληθεί από αυτό. Παρότι οι ίδιες αρχίζουν να αποδέχονται λίγο περισσότερο το Ιράν αλλά έχουν τροφοδοτήσει αυτές τις ανησυχίες της Σαουδικής Αραβίας. Το έχουμε δει ε, στη Σαουδική Αραβία και είναι γνήσιο αυτό. Η άνοδος του Ιράν είναι κάτι που θεωρούν οι Σαουδάραβες ότι είναι σε βάση των δικών τους συμφέροντων, ενώ για πολλές ευρωπαϊκές χώρες υπάρχει ελπίδα ότι όλοι θα έχουν κερδισμένοι από την αλλαγή αυτή, διότι θα μειωθούν οι περιφερειακές εντάσεις. και η αντίδραση που έχουμε στη Σαουδική Αραβία σε σχέση με όλες αυτές τις απειλές ε, ε, θεωρούμενες απειλές έχουμε τον ε, βασιλέα Σαλμάν και τον νεότερο κληρονόμο του μας είπε η Ανίστα σχετικά είναι πιο επιθετική η, η πολιτική πλέον εξωτερική αναζητεί αντιπαράθεση και αυτό ήδη πριν από το Σαλμάν. Υπήρξε απόκληση των πολιτικών, των ευρωπαϊκών και αμερικανών εταίρων πρώτα με τον Μπαχρέιν, η Σαουδική Αραβία και άλλες χώρες της Συμβουλής Συνεργασίας του ΚΟΠ έστειλαν στρατεύματα στον Παχρέν. Ακόμη και αν προσπαθούσε, προσπαθούσαν οι ΥΠΑ να διαπραγματευτούν για μια κυβέρνηση εθνικής ενότητας στη χώρα έπειτα ε, για την ανατροπή του Μόρση. Πάλι ε, αντίδρασαν διαφορετικά οι Σαουδάρβες σε σχέση με τους Αμερικανούς και τους Ευρωπαίους και είπαν ότι από την πλευρά της Σαουδικής Αραβίας αυτές οι χώρες που ήταν στην πίσω αυλή, αν θέλετε, της Σαουδικής Αραβίας ε, είχαν μεγαλύτερη σημασία για αυτούς. Τώρα, ίσως το πιο σημαντικό ζήτημα ήταν η στρατιωτική επέμβαση στην Ιεμένη, που συνιστά μια δραματική αλλαγή στο πλαίσιο ασφάλειας και άμυνας και των σχέσεων με την Σαουδική Αραβία, όπου παραδοσιακά πολλούνταν τα όπλα Σαουδική Αραβία για αμυντικούς αποτρεπτικούς σκοπούς και πολλές φορές υπήρχε μια κοινική αντιμετώπιση μεταξύ τοπικών οικονομολόγων και ε, σχολιαστών στον κόλπο για το βαθμό στον οποίο Σαουδική Αραβία και άλλες χώρες του κόλπου δαπανούσαν χρήματα για την άμυνα. Θα συνδυασμό με τα για την επένδυση χωρίς να φαίνεται ότι υπάρχουν προφανή ωφέλη σε σχέση με τα όπλα. Υπήρχε και μπλοκή τη Σαουδική Αραβία, συμμετοχή τη μάλλον σε ειρηνευτικέ διαδικασίε εκτό των συνόρων, παραδείγματο χάρη ε, στην κατήγεθα τη Ερήμου για την προστασία του Κουβέιτ, αλλά ο πόλεμο τη Εμένη είναι κάτι εντελώ καινούριο στη σύγχρονη ιστορία της Αραβίας. Ναι. επιχείρηση που και από του δικού συμμάχου σε Ηνωμένο Βασίλειο και είπα κυρίω ταυτόχρονα. Saudi Arabia has a marriage emerged υπάρχουν αεροπορικές επιδρομές, περιορισμοί στα λιμένες της Ιεμένης, και αυτό δημιουργεί τεράστια διλήμματα για τις ευρωπαϊκές χώρες σε μία περίοδο που δεν έχουν και τόσο μεγάλη όρεξη είτε για στρατιωτικές επεμβάσεις στη Μέση Ανατολή είτε για ε, χορήγηση ανθρωπιστικής βοήθειας. Βλέπουμε δηλαδή την Ευρώπη αυτή τη στιγμή να είναι διχασμένη. Να έχουμε την ε, Σαουδική Αραβία ε, και άλλες χώρες προσπαθούν να λύσουν τα περιφερειακά προβλήματα, αλλά απ' την άλλη θέλουν να έχουν και λόγο ευρωπαϊκές χώρες. Χωρίς όμως να ασκούν μεγάλη μόχλευση, εφόσον δεν στέλνουν στρατεύματα ή δεν συμμετέχουν με άλλο τρόπο, οικονομικό και άλλο. Είπα κάποια πράγματα για τις ε, σχέσεις, τις αμυντικές, τη φύση αυτών των σχέσεων με κάποιες ευρωπαϊκές χώρες. Πιο σημαντικέ είναι το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία. Το Ηνωμένο Βασίλειο το 2015 είχε τα δύο τρίτα των συμφωνιών εισαγωγών όπλων σε αξία σε σχέση με όλες τις άλλες και εκδόθηκαν 882 άδειες της τάξης των 4 δις ευρώ σε ό,τι αφορά τις παραγγελίες και 11 άδειε μόνο δεν έγιναν δεκτές για λόγους ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Σε μόλις μία περίπτωση η άδεια δεν δόθηκε γιατί θεωρήθηκε ότι μπορεί να υπάρξει εκτροπή σε άλλες ζώνες συγκρούσεων. Παρότι υπάρχουν αναφορές για πώληση όπλων ε, σε χώρες του κόλπου που μετά αυτά τα όπλα βρέθηκαν στη Συρία. Οι συμφωνίες που υπάρχουν λαμβάνει υπόψη να, ε, τις αμυντικές αγοραπολισίες, τις πωλήσει αμυντικού εξοπλισμού και προβλέπουν κάποια κριτήρια. Υποτίθεται ότι πρέπει τα άπλα να πηγαίνουν στην Σαουδική Αραβία και πρέπει να υπάρχει μια πολιτική συνεργασία και κάποια κοινά συμφέροντα. Αλλά προηγουμένη στρατιωτική συνεργασία δεν υπάρχει. Πρόκειται κυρίως για παροχή εξοπλισμού και εκπαίδευσης περισσότερο στατιωτικό προσωπικό στα Δική Αραβία είναι Βρετανοί, 130 περίπου. Και στο Υπουργείο Άμυνας υπάρχουν κάποιοι πολιτικοί αξιωματούχοι, οι οποίοι ασχολούνται με διαγωνισμούς, εκπαίδευση και επικοινωνιακά συστήματα. Επίση αυξάνεται η συνεργασία μεταξύ Γαλλίας και Σαουδικής Αραβίας. Πέρυσι καιροποίησαν την στρατιωτική του συνεργασία, τη σχετική συμφωνία και υπήρξαν δηλώσεις που έλεγαν ότι αυτό γίνεται για την ενίσχυση των αμυντικών διαγωνισμών. Ιδίω ό,τι αφορά το ναυτικό. Η Ισπανία επίσης έχει υπογράψει συμφωνία στρατιωτικής συνεργασία με τη Σαουδική Αραβία από το 2008-2007 για την εκπαίδευση της αεροπορίας, και η Γερμανία επίση, Πολλά όπλα στην ε, Σαουδική Αραβία. Τρίτος μεγαλύτερο αγωγέας ε, γερμανικών όπλων είναι η Σαουδική Αραβία. Βέβαια ακούσαμε πολλά ε, και υπάρχει έντονη συζήτηση για το κατά πόσο θα πρέπει για μένα πολλά όπλα στην Σαουδική Αραβία λόγω των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Στη Γερμανία υπάρχει αυτή έντονη συζήτηση. Βέβαια αυτό που βλέπουμε σε διάφορες χώρες και εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ένα, μια μεγάλη αντίδραση σε σχέση με την Ιεμένη. Αυτή τη στιγμή θα γίνει και μια εξέταση μιας περίπτωσης, μιας ΜΚΟ, γιατί ε, μια, η ΜΚΟ έθεσε θέμα στο δικαστήριο την πώληση όπλων Άρα θα γίνει μια δικαστική εξέταση και έρευνα. Για το μέλλον, ποιες είναι οι μελλοντικές προοπτικές. από το μεγάλο σχέδιο οικονομικών μεταρρυθμίσεων με, όραμα, με ορίζοντα το 2030, κάτι σημαντικό που προέκυψε είναι ότι μέχρι το 2030 η Σαουδική Αραβία θέλει να έχει αυξάσει σημαντικά τις αυτοτικές βιομηχανίες. Αυτή τη στιγμή έχει το 2% μόλις των όπλων της. Με αυτό το νέο ε, σχέδιο, μέσα σε 14 χρόνια, τα μισά, ε, το μισό αμυντικό της εξοπλισμό θα τον εξασφαλίζει με την τόπια παραγωγή. Μάλλον απίθανο να ισχύσει αυτό μέσα στα 14 επόμενα χρόνια. Και αν συμβεί βέβαια, αυτό θα απαιτήσει σημαντικές επενδύσεις και άνοιγμα σε μεταφορά τεχνογνωσίας και τεχνολογίας από ευρωπαϊκές χώρες. Αρκετά αβέβαιο κάτι τέτοιο. Αλλά είναι πολύ ενδιαφέρον γιατί είναι η φιλοδοξία της χώρας αυτής, η επιθυμία της είναι να δημιουργήσει θέσει εργασία στη χώρα. Αλλά έχει και μια βαθύτερη, ένα βαθύτερο νόημα. Ότι δεν θέλει τόσο να εξαρτάται από εξωτερικούς παράγοντες. Γιατί αυτό είναι μακροχρόνιος κίνδυνος. Είναι εντελώ ασαφέ κατά πόσο η Σαουδική επέμβαση στην Ιεμένη αποτελεί μια ένδειξη για αυτά που πρόκειται να έρθουν ή κατά πόσον πρόκειται για μια προσωρινή αντίδραση σε μια προηγούμενη περίοδο μια εξωτερικής πολιτικής η οποία ήταν πολύ προσεκτική. Χρειάζεται πολλή ανάλυση για να θεωρήσει κανεί πως η Εμένη είναι η αρχή μιας νέας, ενός νέου δόγματος του βασιλέα Σαλμάν, το οποίο μπορεί να επεκταθεί και στη Συρία. Η Εμένη δεν ήταν αρκετά επιτυχής ώστε να, αποτελέσει, να αποκτήσει παραδειγματικό ρόλο. Έχουμε πολύ περιορισμένες δημοσκοπήσεις, αλλά από ό,τι φαίνεται ο πόλεμος ήταν αρκετά δημοφιλής στη Σαουδική Αραβία. Το οποίο περιγράφεται συχνά ως πόλεμος αναγκαιότητας για την προστασία γειτονικών αραβικών κυβερνήσεων ε, ε, ενάντια σε πραξικοπήματα. αλλά υπό το πρίσμα της εγχώριας λιτότητας είναι όλο και λιγότερο πιθανό να διατηρηθεί αυτή η στάση. Και έτσι είναι σχετικά πιθανό η Σαουδική Αραβία να αναλάβει την ηγεσία, τη στρατηγική ηγεσία της Μέσης Ανατολής. Είναι πιο πιθανό να υποθεί πως εξωθηθήκαμε στην κατάσταση αυτή επειδή οι παραδοσιακοί σύμμαχοι μας από τη Δύση μας άφησαν μόνους μας. Τέλος, όσον αφορά τις μελλοντικέ προοπτικές, πιθανώς η, εκεί που θα διχαστούν τα πνεύματα είναι το Ιράν. Πολλά ευρωπαϊκά κράτη-μέλη θα ήθελαν πάρα πολύ να, επεκτείνουν τις οικονομικές του σχέσεις με το Ιράν, ενώ η, η Σαουδική Αραβία το θεωρεί ως την κύρια απειλή και θεωρεί τη χώρα αυτή σε μεγάλο βαθμό υπεύθυνη για την άνοδο του ISIS. Μπορούμε να βαθύνουμε σε αυτό περισσότερο στη συζήτηση. Αλλά ο παράγοντας του Ιράν είναι καθοριστικός για το φαινόμενο των πολέμων διατυπροσώπων στην περιοχή, όπως φαίνεται στη Συρία. Ωστόσο τα ευρωπαϊκά κράτη-μέλη θα πρέπει να θεωρούν πιθανά όλα τα σενάρια και να τα εξετάσουν κατά τη σύσπηξη των εξοπλιστικών του σχέσεων με τη Σαουδική Αραβία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. κυρίες, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την τόσο ολοκληρωμένη και τόσο ενδιαφέρουσα παρουσίαση. Δεν υπάρχουν τόσο πολλά μέλη εδώ, λόγω διάφορων περιορισμών, αλλά πιστεύω πως μπορούμε να προχωρήσουμε σε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Μαρακιούρα. κυρία Βαλέρο. Συγγνώμη, κατά κάποιο τρόπο μπερδεύτηκε η σειρά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα αυτά που μας είπατε εδώ. Πιστεύω πως ήταν πολύ, είχε πολύ ενδιαφέρον να σας ακούσουμε. Ακούσαμε πολλά για την εξαγωγή όπλων. Είμαι από τη Σουηδία, όπου από ό,τι ξέρετε υπήρξε ένα μεγάλο σκάνδαλο. Όταν ο κόσμος αντιλήφθηκε πως προσπαθούσαμε να βοηθήσουμε τους Σαουδάραβες να δημιουργήσουν μια βιομηχανία όπλων χωρίς κανείς να το ξέρει. Όλα έγιναν μυστικά. Φυσικά και πιστέψαμε πως αυτό είναι αντίθετο με το Σουηδικό νόμο. Αλλά αντιληφθήκαμε επίσης πως έχουμε ένα μνημόνιο κατανόησης με τους Σαουδάραβες το οποίο και πέρυσι δεν ανανεώσαμε. Γι' αυτό και το μνημόνιο αυτό έχασε την ισχύ του. Οι σχέσεις με τη Σαουδική Αραβία σε άλλα θέματα που δεν, που δεν σχετίζονται με την άμυνα υπάρχουν ακόμα, αλλά όσον αφορά τις εξαγωγές όπλων κτλ. ένας από τους κύριους λόγους που έχουν ταραχθεί τόσο οι άνθρωποι στη χώρα μου είναι τα ζήτημα πέραν των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είναι μέσα στα ανθρώπινα δικαιώματα κυρίως τα δικαιώματα των γυναικών. Και φυσικά υπάρχει μια κοινή θέση, έχουμε έγγραφα σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και σχετικές εκθέσεις, αλλά τα δικαιώματα των γυναικών δεν είναι τόσο ισχυρά και μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε για να σταματήσουμε τις εξαγωγές προς τη Σαουδική Αραβία. Θα ήθελα λοιπόν να ακούσω επειδή θίξαμε τόσο πολλά τις εξαγωγές όπλων, έχουμε τον πόλεμο στην Ιεμένη, εμείς από το Κοινοβούλιο θέλαμε ένα εμπάργο στις εξαγωγές όπλων προς την Ιεμένη, συγγνώμη, προς τη Σαουδική Αραβία, λόγω της Ιεμένης. Συμβαίνουν λοιπόν πάρα πολλά πράγματα. Αναρωτιέμαι λοιπόν κατά πόσον επηρεάζει αυτό τους Σαουδάραβες. Επειδή παραδείγματο χάρη ξέρω πως έχουν πλέον δημοτικές εκλογές στις οποίες μπορούν να συμμετάσχουν και οι γυναίκες. Αυτό οφείλεται στην πίεση που προέρχεται από τους εταίρους της χώρας στην Ευρώπη. Ελπίζω τουλάχιστον να έχει φτάσει μας κάποιον αντίκτυπο, αλλά θα ήθελα να ακούσω από εσάς κατά πόσον συντρέχει αυτό. Αυτά που εμείς κάνουμε έχουν κάποιον αντίκτυπο σε αυτά που συμβαίνουν στην κοινωνία των πολιτών εκεί, ώστε να πέθουν αλλαγές. Θα ήθελα επίση να θέσω μια ερώτηση, αλλά θέλω και ένα σχόλιο από την κυρία Λεβαλουά, το εργαστήριο αυτό προετοιμάστηκε για να ασχοληθούμε με ζητήματα ασφάλειας και άμυνας. Ασφαλώς και υπάρχουν συγκεκριμένες πτυχές ενός εμπάργου, εμπάργου στις εξαγωγές όπλων και βρισκόμαστε σε μια πολύ ευαίσθητη κατάσταση καθώς το εργαστήριο αυτό συγκλήθηκε ξεχωριστά εντός της ΣΕΝΤΕ και δεν θα έπρεπε να επισέλθει πολύ βαθιά στο αντικείμενο άλλων υποεπιτροπών. Είναι φυσικά δύσκολο να αποφύγουμε ορισμένες άλλοι επικαλύψεις όσον αφορά κάποιες πτυχές ή ζητήματα. Ωστόσο θα προτιμούσα να εστιάσουμε σε ζητήματα ασφάλειας. Είχαμε μια πολύ καλή παρουσίαση. Επειδή υπάρχουν πολλές προτεραιότητες ασφάλειας και άμυνας και πολλές ανησυχίες σχετικά με αυτό που πρέπει να συζητηθούν επίσης. Με γνώση αυτού θα ήθελα να γνωρίσω και τις δύο προσκεκλημένες να μας παρουσιάσουν σύντομα τις εντάσεις μεταξύ Σουνιτών και Σιητών στην περιοχή. Πόσο σημαντικές θεωρείτε πως είναι αυτές οι εντάσεις. Θα έλεγα σε περιοχές σημαντικών συγκρούσεων, ιδίω στη Συρία, το Λίβανο, το Ιράκ, αλλά επίσης στην Ιεμένη σε κάποιο βαθμό. Γνωρίζουμε τους σημαντικούς παράγοντες, τους σημαντικούς δρόντες και τις δυνάμεις που δραστηριοποιούνται σε αυτό το πλαίσιο. Γνωρίζουμε τις δύο ομάδες του Ισλάμ. Ωστόσο θα ήθελα να ακούσω για τις δυναμικές που υπάρχουν με το ιστορικό υπόβαθρο που υπάρχει. Ο κύριος Λόπες, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα μια σύντομη δήλωση και μετά η ερώτηση, η οποία έχει να κάνει με το θέμα. Ελπίζω, με συγχωρείτε πρώτα απ' όλα που καθυστέρησα, δεν παρακολούθησα όλη την συζήτηση, ίσως να το είπατε ήδη, αλλά εδώ έχουμε ένα πάνελ με θέμα της Σαουδική Αραβία. Δεν μπορούμε όμως να δούμε το θέμα αυτό χωρίς να δούμε και το Ιράν σχετικά. Ελπίζω να είμαστε τόσο σαφείς και διαφανείς με το Ιράν, όπως θα πρέπει να είμαστε και με τη Σαουδική Αραβία και για τους εξοπλισμούς και για όλα. Υπάρχει μια ε, τάση στην ε, Ευρωπαϊκή Αριστερά να είμαστε κάπως επιότεροι με το Ιράν. Όποιοι και να είναι οι λόγοι, μοναρχία, ιστορικοί λόγοι, δεν ξέρω ποιοι είναι, το μόνο που ρωτώ είναι αν πρέπει να παίξει κάποιο ρόλο η Ευρώπη και ίσως κάποια στιγμή θα κληθούμε να το κάνουμε αυτό και ε, θα πρέπει να έχουμε τότε την τόλμη κάτι να κάνουμε. Ε, αν το κάνουμε λοιπόν αυτό, θα πρέπει να έχουμε μια ισόρροπη προσέγγιση στην περιοχή. Διότι υπάρχουν πολλοί παράγοντε εδώ, όχι μόνο η Σαουδική Αραβία και το Ιράν και τα αντικρώμενα συμφέροντά του στην περιοχή. Υπάρχει τώρα και παρουσία άλλων παραγόντων, όπω τη Συρία ή η Ρωσία. Και το πρόβλημα δεν είναι η Συρία, είναι λόγω χάρη η Αίγυπτος. Η Αίγυπτος έχει στρατηγική σημασία. Η σχέση της Σαουδικής Αραβίας με την Αίγυπτο και αυτή είναι στρατηγική. Τι νομίζετε θα συμβεί λοιπόν εάν η Ρωσία πλησιάσει περισσότερο την Αίγυπτο. Τι αλλαγές ε, θα προκαλέσει, μάλλον οι αλλαγές στις, σχέσεις, στις στρατηγικές σχέσεις Αιγύπτου-Σαουδικής Αραβίας, πώς θα επηρεαστούν. Πρόεδρος, ναι, Αναφέρθηκε σίγουρα αυτό στις προηγούμενες ε, παρουσιάσεις, αλλά αξίζει να το δούμε περαιτέρω. Κυρίες μου, έχετε το λόγο. Πρώτα απ' όλα η κυρία Λεβαλουά και μετά η κυρία Κίνεμον. Ευχαριστώ για τις διάφορες ερωτήσεις. Θα προσπαθήσω να απαντήσω. Να ξεκινήσω από την τελευταία. Διότι όντω υπάρχει σημαντική σχέση αυτή τη στιγμή και νέε επαφέ μεταξύ Αιγύπτου και Ρωσία. Βλέπουμε ότι ο Πούτιν Όντω θέλει να ξανααναθερμάνει τις σχέσεις με την Αίγυπτο. Σχέσεις Αιγύπτου-Ρωσίας υπήρχαν ε, από λόγους ιστορικούς. Ε, η συμμαχία με την Ουάσογκτο βεβαίως τις κατήργησε, αλλά σήμερα βρισκόμαστε σε μια φάση που η Ρωσία προσπαθεί να ε, ξανακάνει σε την παρουσία της όλη την περιοχή. Με κάποια επιτεύγματα σαφή. Το βλέπουμε και στην περίπτωση τη Σαουδική Αραβία με σχέσει που έχουν αναθερμανθεί με τρόπο αρκετά ε, αξιοσημείωτο μεταξύ Μόσχα και Ριάντα, Μόσχα και Καΐρου. Και όλα αυτά είναι ένα νέο στοιχείο που πρέπει να λάβουμε υπόψη ε, στην ε, περιοχή στο τι συμβαίνει στην περιοχή, διότι η Ρωσία παίζει ένα ρόλο ε, στην ε, Συρία, βλέπουμε και πόσο σοβαρή εμπλοκή έχει, αλλά βλέπουμε και την διάθεση της Ρωσίας να είναι έντονη η παρουσία της και πραγματικά και εκεί να μπορεί να προσφέρει αμυντικό εξοπλισμό, να πουλάει όπλα ε, και θέλει να είναι μια από τις βασικότερες πηγές ανεφοδιασμού. Βλέπουμε τι γίνεται με την, ε, στη σχέση με την Αίγυπτο, ε, βλέπουμε τι γίνεται και με τη Σαουδική Αραβία. Είναι πολύ σημαντικά αυτά και θα πρέπει εμεί οι Ευρωπαίοι σε κάθε περίπτωση να τα σκεφτούμε. Να τα σκεφτούμε στο πώ προσεγγίζουμε αυτή τη γεωγραφική περιοχή και την ασφάλεια εκεί. Για να δούμε και εμεί ποια είναι η θέση μα ω Ευρωπαίοι Διότι θα πρέπει να συνδυαστούμε με του Αμερικανού και του Ρώσους που έχουν μια σημαντική παρουσία εκεί, αλλά υπάρχουν διαφορέ μεταξύ του. Η Ρωσία θέλει να διεκδικήσει τη θέση της, να έχει τα απαραίτητα μέσα και να υψώσει το αναστημά τη απέναντι στην Αμερική, που θα αλλάξει ίσω γιατί έχουν και εκλογέ, αλλά τα τελευταία χρόνια δεν θέλει αμέσω να διαχειρίζεται, ε, θέλει να, να έχει τον έλεγχο βέβαια, αλλά δεν θέλει αμέσω να διαχειρίζεται τα πράγματα εκεί και αφήνει κάποια θέση στη Ρωσία. Στη Ρωσία που είναι αποφασισμένη να προχωρήσει και να είναι αποτελεσματική στη δράση τη και να είναι πραγματικό εταίρο για τι χώρε με τι οποίε είναι από τι σχέσει. Αυτό θέτει ένα ερώτημα για τον ρόλο των Αμερικανών και το πόσο αξιόπιστη είναι αυτή η συμμαχία πλέον. Πέραν αυτών, σημαντικό, τα τελευταία χρόνια ενδιαφέρον μάλλον τα τελευταία χρόνια είναι πέραν τη ρασία που επανέρχεται στο προσκήνιο, αυτό που βλέπουμε με σαφήνεια να σχηματίζεται, είναι να έχουμε περισσότερε περιφερειακέ δυνάμει στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή. Δηλαδή τα προηγούμενα χρόνια με τι αραβικέ επαναστάσει ήταν κυρίω οι Αμερικανοί και οι δυτικέ δυνάμει που ε, έσερναν το χορό, για να το πω έτσι, στην περιοχή. Σήμερα βλέπουμε περιφερειακέ δυνάμει να, ε, καταλαμβάνουν τη θέση που του αρμόζει όχι πλέον ε, χωρίς την αιγίδα των ε, ε, εξωτερικών, των διεθνών τους νονών, για να το πω έτσι, των προστατών τους, αλλά Τώρα, η αλλαγή που βλέπουμε σε αυτή τη γεωγραφική περιοχή είναι ότι οι περιφερειακές αυτές δυνάμεις αντιλαμβάνονται το ρόλο που θέλουν να διαδραματίσουν και την συνείδηση ότι έχουν ένα πραγματικό ρόλο να διαδραματίσουν. όπως είπα, ε, με τους προστατές και με το Ιράν να προστατεί. Αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη στην όλη μας ανάλυση για να καταλάβουμε πώς εμείς μπορούμε να τοποθετηθούμε σε σχέση με αυτά τα νέα ε, στοιχεία με το γεγονός ότι υπάρχουν νέες περιφερειακές δυνάμεις που αρχίζουν να ε, αυτονομούνται και που ε, αρχίζουν να σχεδιάζουν τι πολιτικέ τους με βάση τα δικά του συμφέροντα και όχι μόνο να δέχονται τις ε, πολιτικές που τους επιβάλλουν οι νονοί από τις δυτικέ δυνάμεις, οι προστάτες του δηλαδή, όχι μόνο οι Αμερικανοί αλλά και οι Ευρωπαίοι και το καταξύ. λίγα λόγια για του Σουνίτε και του Σιήτες εδώ τι γίνεται με την ε, αναρχία στις δύο θρησκευτικέ ομάδες και τα θρησκευτικά δόματα στα οποία ε, δίνεται τόση έμφαση. Εγώ ανήκω σε αυτούς που θεωρούν ότι το να μιλάμε για θρησκεία βεβαίως είναι ένα στοιχείο που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη, αλλά αυτά είναι ε, σκέψεις στρατηγικές και γεωπολιτικές που ξεπερνούν τα όρια των θρησκειών. Δεν πρέπει να αυταπατώμεθα. Δεν νομίζω ότι πρέπει να βλέπουμε την περιοχή αυτή και να τη μελετάμε υπό το πρίσμα αυτών των δύο θρησκευτικών ομάδων, Σουνιτών και Σιτών, που αντιπαρατήθενται. Δεν αντιπαρατήθενται μόνο για τα θέματα τη θρησκεία, κυρίω έρχονται σε σύγκρουση για θέματα πολιτικά και θέματα γεωπολιτικά μάλιστα. Νομίζω λοιπόν ότι δεν πρέπει να ε, αυταπατώμεθα, όπω είπα. Δεν λέω ότι η θρησκεία δεν έχει τη σημασία τη. Βεβαίω θα ήταν ανοησία να βεβαιώσει κανεί κάτι τέτοιο. Όμως να μην περιοριζόμαστε στο να λέμε ότι οι Ιρανοί θέλουν θέλουν ε, να φάνε τους ε, Σαουδάραβες ε, Σουνίτες ή αντιστρόφως γιατί το πρόβλημα δεν είναι αυτό είναι ότι θέλουν βεβαίω κάποιοι να διατηρήσουν την ομοποίησή του στου ιερού θρησκευτικού χώρου. Αυτό είναι μια θρησκευτική διεκδικήση και είναι πραγματική και χειροπιαστή. Υπάρχει όμω πάνω απ' όλα πολιτικό ζήτημα. Μην μπερδευόμαστε και το προσεγγίζουμε αλλιώ. Γιατί αλλιώ δεν θα καταλαβαίνουμε τίποτα και θα χάσουμε και τη δυνατότητα να διαχειριστούμε, να αξιολογήσουμε και να βρούμε τι σωστέ αποκρίσει σε αυτά τα ζητήματα. Θα μου πείτε βεβαίω, αν δεν κανεί την κατάσταση στη Συρία, πραγματικά καταλαβαίνει ότι έχουμε να κάνουμε με μια αντιπαράθεση Σουνιτών σιτών. Όχι, πάνω απ' όλα μιλάμε για ένα πόλεμο, τον οποίο τον ε, διεξάγει ένα μέρο ε, του πληθυσμού κατά του απολυταρχικού καθεστώτο και η έναρξη τη επανάσταση στη Συρία δεν είχε καμία σχέση με την έναρξη αλαβητών και Σουνιτών, σιτών και Σουνιτών. Ε, είναι σφάλματα που προσεγγίζει κανεί έτσι. Τώρα, έτσι. Τώρα το να προσπαθεί κανείς να δει τον πόλεμο μέσω από πρίσμα ε, θρησκευτικό αποκλειστικά και μόνο, είναι και αυτό μια επιλογή. Αλλά θα πρέπει να είναι κανεί πολύ επιφυλακτικό, ιδιαίτερα συνετό και να μην σφάλει στον τρόπο που προσεγγίζει τα πράγματα. Και με ένα τελευταίο σχόλιο για το ρόλο των γυναικών στην κοινωνία. Στην ε, Σαουδική Αραβία πήγα πριν από λίγου μήνε και πραγματικά ξεπλάγει όταν είδα ότι υπάρχει πραγματικό κίνημα στους κόλπους της αοδικής κοινωνίας και ότι οι γυναικές αρχίζουν να διδραματίζουν όλο ένα και σημαντικότερο ρόλο. Ένα ρόλο κυρίως από τα στρώματα των καλλιεργημένων, των μορφωμένων γυναικών της ε, κοινωνίας της Σαουδικής Αραβίας, του πρώτου επίπεδου θα έλεγα, του ανώτερου επίπεδου, αυτές οι γυναίκες θέλουν κάπως τα πράγματα να πάρουν μπρος και να αρχίσουν να κινούνται και για αυτές. Όμως ε, βλέπουμε αυτές οι γυναίκες που έχουν επιχειρήσεις, που είναι μορφωμένες και καλλιεργημένε, καταλαβαίνουν ότι τα πράγματα πρέπει να αρχίσουν να κινούνται εκ των έσω. Με αυτήν την αυτοεικόνα ότι η εξωτερική πίεση που πρέπει να αντιμετωπίσουν με τρόπο διακριτικό για να μην διαταράξουν τι ισορροπίε και τη βασιλική οικογένεια που δεν ανέχεται με τίποτα την οποιαδήποτε εξωτερική παρέμβαση. Τέλο πάντων, προσπαθούν να συζητήσουν και να διαπραγματευτούν με του ηθήνοντε τη Σαουδική Αραβία, μα και κάπω πάρουν μπροστά πράγματα στη Σαουδική κοινωνία, αλλά με τρόπο διακριτικό. Χωρί αυτό να ε, γίνεται θέμα και να προβάλλεται, γιατί αυτό μπορεί να δυσκολέψει τα πράγματα. Οι συζητήσει και αυτέ οι πιέσει που ασκούνται λοιπόν είναι χρήσιμε, μπορεί να φέρουν αποτέλεσμα, αλλά πρέπει κανεί να πηγαίνει ε, ψηλαφώντα και πολύ προσεκτικά, ώστε να μην ε, ε, η κοινωνία και ξανακλείσει στο καβούκι τη πρέπει να έχει την αίσθηση ότι δεν υπάρχουν εξωτερικέ πιέσει. Και έτσι μπορεί και να ανοιχτεί λίγο και παραπάνω. Πάντω υπάρχουν κάποιε συνεννοήσει, κάποιε πιέσει, με πάρα πολύ σύνεση βέβαια, για να είναι αποτελεσματικέ εν τέλει και όλα αυτά με ε, την ε, ελπίδα ότι θα μπορεί να υπάρξει μια εσωτερική εξέλιξη. Πρόεδρο, ευχαριστούμε κυρία Κίνεμοντ. Ευχαριστώ. Να επανέλθω σε αυτό το θέμα των εξωτερικών πιέσεων και ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδίω σε σχέση με τι εξαγωγέ όπλων. Υπάρχει πραγματική δυσκολία να αξιολογήσει κανείς τι είναι αποτέλεσμα εξωτερική πίεση. Συνήθως, αν είναι αποτελεσματική η εξωτερική πίεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα, αυτό συμβαίνει μόνο αν υπάρχει και στο εσωτερικό επίπεδο ε, ένας πυρήνας που θέλει να προχωρήσουν ε, αυτά τα ανθρώπινα δικαιώματα, να υπάρχει σεβασμός τους. Αλλά για κάποιες χώρες που είναι πολύ κοντά στη Σαουδική Αραβία, για την Ευρώπη μιλάω, ε, κάποιες από αυτές τις χώρες ε, επιχειρηματολογούν ότι με την παροχή όπλων έχουν και ένα μέσο ε, άσκησης επιρροής. Φυσικά δεν είναι αυτή ο κινητήριος μοχλός, γιατί εδώ μιλάμε και για πολύ χρήμα, αλλά είναι ένα επιχείρημα που ακούγεται από ορισμένους, ότι δηλαδή μια χώρα η οποία δίνει όπλα μπορεί επίσης να απαιτήσει καλύτερη εποπτεία και έλεγχο ό,τι αφορά την τήρηση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, μπορεί να στάει πληροφορίες για τα συστήματα που υπάρχουν για τη διερεύνηση υποθέσεων, περιπτώσεων καταχρήσεων κτλ. Αυτό μπορεί να έχει κάποιο νόημα, αλλά αν και μέσα στο αμυντικό establishment της Σαουδική Αραβία υπάρχει ένας ε, πυρήνας που θεωρεί ότι είναι στρατηγικό κόστος τα θύματα μεταξύ των αμάχων. Οι διπλωμάτες δηλαδή να πούν ότι δεν θέλουμε να σκοτώνουμε αμάχους. Οι άμαχοι βέβαια πεθαίνουν και αυτοί, ε, όπως και στο Ιράκ, είναι μια απώλεια, αλλά δεν είναι στόχος μας, δεν θέλουμε να συμβαίνει αυτό. ή μπορεί θα υπάρχουν περιπτώσεις που θεωρεί ότι αυτοί οι περιορισμοί είναι τεχνητοί, είναι υποκριτικοί, δηλαδή ότι τους ε, κατηγορούν ε, και τους καταγγέλουν για παραβιάσεις των δικαιωμάτων του πολύ περισσότερο από άλλες χώρες για τις χώρες που παρέχουν τα όπλα επίσης υπάρχει ο κίνδυνος ότι όσο πιο πολύ κανείς συμμετέχει, δηλαδή δεν παρέχει μόνο όπλα, αλλά και την εποπτεία και βοηθά με τα συστήματα, τότε μπαίνει και πιο μέσα στην ίδια την σύγκρουση. Όπως στην περίπτωση του νομού Βασιλείου, για παράδειγμα, που πολλοί οι θεωρούν ότι είναι πλέον ένα εμπλεκόμενο μέρος αυτή τη σύγκρουση και όχι ένας διαμεσολαβητής ή παρατηρητής για τις εντάσεις μεταξύ Σιητών Σουνιτών. Συμφωνώ ότι η γεωπολιτική είναι η λόγη των εντάσεων και αυτό μπορούμε να το εξηγήσουμε γιατί από 14 αιώνε βλέπουμε αυτές τις εντάσεις. Το θέμα που μας ανησυχεί είναι ότι οι περισσότεροι στο Ιράν και στη Σαουδική Αραβία είναι νέοι κάτω των 30. Και όσο καιρό έχουν πολιτική συνδεσία, αν έχουν βέβαια, αυτό που βλέπουν στις ειδήσει είναι αυτές οι, οι εντάσεις και οι συγκρούσεις μεταξύ διαφόρων φιλών, φατριών. Άρα θεωρούν ότι αυτό είναι πιο σημαντικό, οι φατρίες, οι φιλές και οι κοινότητες που ανήκουν. Πολύ πιο σημαντικό για αυτούς σε σχέση με τις παλιότερες γενιές. Και αυτό είναι ένα δυσεπίλητο πρόβλημα. Οι ευρωπαϊκές χώρες όμως δεν θα πρέπει να το δουν στο εσωτερικό ε, μόνο πρόβλημα, σε εσωτερική αντιπαράθεση. Είναι γεωπολιτική σημασία και έχω συνεισφέρει και αυτή. Λοιπόν, ένα σημαντικό ερώτημα ήταν για τη Ρωσία και την Αίγυπτο. Ήδη το είδαμε να ξεκινά αν θέλετε, αλλά η Αίγυπτος σε μεγάλο βαθμό χρησιμοποιεί τη Ρωσία για να στείλει ένα μήνυμα στη ΣΥΠΑ ότι έχει εναλλακτικέ Υπάρχει επίσης προσέγγιση Αιγυπτου-Κίνας για επενδύσεις βέβαια και όχι τόσο για την άμυνα. Δεν ξέρουμε τώρα αν θα μπορούσε να αρκεί ε, η Ρωσία και η Κίνα αν απομακρυνθεί εκτός από την ε, ΣΥΠΑ. Τώρα δεν ξέρω η Ρωσία πώς μπορεί να επηρεάσει, μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τις σχέσεις με την ε, Σαουδική Αραβία. Υπάρχει και έλλειψη ίσως ε, χρημάτων ε, από ανθρωπιστική βοήθεια που δημιουργεί κάποια προβλήματα. Σαουδική Αραβία το δυνάμει σαν την Κίνα, σαν τη Ρωσία θα διαδραματίζουν φαίνεται πάντως στο μέλλον περισσότερο ρόλο στην περιοχή και οι δυνάμει οι, οι θα προσπαθούν να πάρουν ε, με το μέρος τους ή να παίξουν τα διεθνών δυνάμεων, για να προσερετεριστούν αυτές και δεν θα είναι τόσο ψυχροπολεμική, αν θέλετε, κατάσταση. Ευχαριστώ. Πολύ ενδιαφέρουσα ανταλλαγή απόψεων, λέει η πρόεδρος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Υπάρχει κάποιος που να θέλει το λόγο. Θα συνεχίσουμε λοιπόν με την ημερήσια διάταξη. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα μια τέτοια επισκόπηση της περιοχής όταν έχουμε σίγουρα μεγάλες αλλαγές στο σύστημα εξουσίας και μεγάλες ανησυχίες όσον αφορά σημαντικούς δρόμους. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά για μας να τα γνωρίζουμε, να τα μαθαίνουμε. Ήταν μια πολύ ολοκληρωμένη και ενδιαφέρουσα επισκόπηση και θα ήθελα τώρα και προσωπικά να μάθω κατά πόσον υπάρχουν ενδείξεις για αυτό που παρατηρούμε στην Ευρώπη όσον αφορά τη δραστηριοποίηση ριζοσπαστικών ή ριζοσπαστικοποιημένων οργανώσεων όσον αφορά τη στρατηγική επικοινωνία κατά πόσον υπάρχουν ενδείξεις για έναν πόλεμο πληροφοριών στο διαδίκτυο, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης στην περιοχή. Κατά πόσον είναι κάτι τέτοιο ορατό. Μπορείτε να αναφερθείτε στο ζήτημα αυτό και στο κατά πόσον νέοι ή ανανεωμένοι δρόντες όπως η ανανεωμενοι δρομτες οπως φαίνονται επίσης σε αυτό σε αυτόν πόλεμο πληροφοριών. Ακούστε, σίγουρα ο ρόλος είναι πολύ σημαντικός. Ε, ένα αποκαλυπτικό σημάδι είναι ότι όλα τα διεθνή μέσα ενημέρωσης σήμερα ε, έχουν κανάλια που μεταδίδουν στα αραβικά, ρωσικά κανάλια, αγγλικά, γαλλικά, ιρανικά, κινέζικα τουρκικά. Άρα υπάρχει και ένας πραγματικός πόλεμος και μια πραγματική βούληση από τις περιφερειακές και διεθνείς δυνάμεις να καταλάβουν και αυτό το έδαφος της επικοινωνίας και η Ρωσία για παράδειγμα δραστηριοποιείται ενεργά στον τομέα αυτό σε σχέση με τις διάφορες συγκρούσεις και εδώ βλέπουμε πραγματικούς πολέμους από όλου τους ε, παρόντες φορείς. Και όπως έλεγα πριν, βλέπουμε ότι όλες οι περιφερειακές δυνάμεις έχουν επενδύσει με αυτό. Ακριβώς για να μπορούν να έχουν επιρροή και για να μπορεί να περνάει το μήνυμα, να περνούν ιδέες και για να γίνει αντιληπτή αυτή η περιοχή ε, με όλες τις ε, με όλα τα προβλήματα που βλέπουμε και έχουμε την αντίληψη ασφάλειας, την αντίληψη της άμυνας για όλους τους φορείς, όλοι οι σκοποί ε, είναι μάλλον όλα τα μέσα είναι καλά για την επίτευξη του σκοπού. Κυρία Κίνιν είναι παράγοντας πράγματι. Η Ρωσία, για παράδειγμα, προσπαθεί να έχει μια αφήγηση αντιπεριαλιστική για τη Συρία λέγοντας ότι οι ΙΠΑ προσπαθούν να καταλάβουν τη Μέση Ανατολή, παρότι η Ρωσία παίζει και αυτή το ρόλο της εκεί. Και για τους περιφερειακούς παράγοντες, Ιράν κτλ. Και η Αραβία έχουν επενδύσει στην προπαγάνδα, δορυφορικούς ε, τηλεοπτικούς σταθμούς, ε, ε, ένα πόλεμο μηντιακό και φυσικά πολλές φορές αυτό γίνεται ένα όπλο. Και αυτό είναι πολύ επικίνδυνο. Κύριος που ρώτησε κάτι το Ιράν. Νομίζω ότι είναι σχετικό. Γιατί εδώ φαίνεται Υπάρχει μια μεγάλη, ένα μεγάλο χάσμα μεταξύ ε, της αφήξης εδώ στην Ευρώπη και της πραγματικότητας. Ενώ ακούγονται πολλά καλά λόγια για το Ιράν. Οι σχέσεις όμως στην πράξη δεν είναι τόσο ε, καλές θερμές αν θέλετε. Και το Ιράν επίσης πόρο απέχει του να έχει ακόμη κάποια αμυντική συνεργασία. Υπάρχει όμως μια σφαλμή αντίληψη ε, στη Σαουδική Αραβία ότι ε, στο Ιράν συγχωρούνται τα πάντα, αλλά στη Σαουδική Αραβία τίποτα. Και Ευρωπαίοι που προσπαθούν να ασκήσουν πιέσει στη Σαουδική Αραβία για θέματα όπως ανθρωπιστικό δίκαιο και δίκαιο πολέμου κτλ. Αυτό πρέπει να είναι σαφές, να μπει σε ένα πλαίσιο για να καταλάβει η Σαουδική Αραβία ότι για αυτήν δεν ισχύουν άλλα μέτρα σταθμά θα ήθελα να ήθελα αυτό το εργαστήριο να μην φανεί σαν μια μονομερή εξέταση του ζητήματος. Θα πρέπει να ασχοληθούμε επίσης με ζητήματα ασφάλειας και άμυνας και μάλιστα παγκόσμιας ασφάλειας και να αξιολογήσουμε τις πολιτικές του Ιράν και να καταρτήσουμε μια επισκόπηση της εκπλήρωσης της συμφωνίας. Θέλουμε να κάνουμε μια επισκόπηση δηλαδή των παγκόσμιων απειλών στην περιοχή τόσο στη Μέση Ανατολή όσο και στη Βορειοαφρική και πάμε θέμα με θέμα και είμαι πολύ ικανοποιημένη με το αποτέλεσμα του εργαστηρίου αυτό, αυτού. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τις δύο ερευνήτριες και τη, για την τόσο αμερόληπτη, τόσο με τόση βαθιά γνώση, εκ των έσω εικόνα της παρουσίασης που μας έδωσαν σχετικά με τις συγκρούσεις στην περιοχή. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Κλείστο λίγο. Please stay, we have second point of our στο δεύτερο τμήμα. Just two minutes for... Λίγα λεπτά λεπτά για να ξανακαθίσουμε στο Προεδρείο. Το Υπότιτλοι AUTHORWAVE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

Ladies Κυρίες και κύριοι, παρακαλώ καθίστε. Να ξεκινήσουμε. Το τελευταίο βασικό σημείο, το τελευταίο μας μάλλον σημείο στην Μέση διάταξη της Επιτροπής ΣΕΝΤΕ για σήμερα, εξαιρετικά ενδιαφέρον, παρόλο που θα γνωρίζετε ότι υπάρχουν κάποιες δυσκολίες δημόσια η συνεδρίασή μας και θα συζητηθεί σίγουρα και στην κοινή γνώμη το θέμα αυτό σε άλλες περιπτώσεις. Εδώ θα μιλήσουμε για την απειλή από χημικά, πυρηνικά, ε, βιολογικά ε, όπλα ε, κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ήθελα να παρουσιάσω τους δύο εξέχοντες προσκεκλημένους μας. Πρώτα απ' όλα ο κύριος Μπρούνο Ντιπρέ της ΑΕΔ Το αντικείμενό του είναι η πολιτική ασφάλεια και η πολιτική διαστήματο και έχουμε και εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή από τη Γενική Διεύθυνση Home. Είναι μεγάλη μου χαρά και τιμή να παρουσιάσω τον κύριο Ζόρζε Μανουέλ Μπέν του Σίλβα και θα ακούσουμε τις παρουσιάσεις τους. Να ξεκινήσουμε με την παρουσίαση της ΕΕ και μετά και να δούμε ε, τις απόψεις του κυρίου Ντιπρέ εάν ε, θέλει για τα θέματα των χημικών όπλων και μετά θα ακούσουμε τον κύριο Μπέντο Σίβλα. Σίλβα. Mrs. Chair. Κυρία Πρόεδρε και κεκριμένα μέλη, αγαπητοί συναδελφοί Επιτρέψτε μου πρώτα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στην Επιτροπή αυτή και σε σας κυρία Πρόεδρε για τη δυνατότητα που δίνεται στην ΕΕΔ να μιλήσει για χημικά, βιολογικά, ραδιοπυρηνικά όπλα και εκρηκτικά που αποτελούν μια πρόκληση για την ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρώτα απ' όλα θα αναφερθώ στον κίνδυνο, στη συνέχεια στο πόσο προετοιμασμένη είναι η διεθνής κοινότητα και δεύτερον και τρίτον ποια μέτρα παίρνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τη βελτίωση της πρόληψης στον ευαίσθητο τομέα αυτό. Πρώτα απ' όλα, η Ευρωπαϊκή Ένωση ανησυχεί βαθιά για τέσσερις κύριες προκλήσεις ασφάλειας οι οποίες ενέχουν όλες μια μεγάλη πιθανότητα χημικής, βιολογικής, ραδιοπυρηνικής απειλή. Το πρώτο είναι η κλιματική αλλαγή, το δεύτερο η τρομοκρατία, τρίτον η ενεργειακή ασφάλεια και τέταρτον η βιοτεχνολογία. Κάθε ένα από τα θέματα αυτά περιέχει σίγουρα απειλές από χημικούς, βιολογικούς και ραδιοπυρηνικούς παράγοντες. Αλλά όλοι αυτοί οι παράγοντες μαζί μπορεί να είναι καταστροφικοί. Α φανταστούμε παραδείγματο χάρη μια βιολογική απειλή σε μια περιοχή που πλήττεται από την κλιματική αλλαγή. Κανείς σήμερα δεν μπορεί να προβλέψει τις καταστροφικές συνέπειες και το εύρος των συνεπειών μιας τέτοιας εγκληματικής πράξης. Ωστόσο, κάτι είναι σίγουρο. Δεν θα περιοριστεί στο, σε ένα κράτος ή σε μια περιοχή. Δεύτερον, πόσο καλά προετοιμασμένη είναι η διεθνής κοινότητα. Ο τρόπος με τον οποίο η διεθνής κοινότητα αντιμετώπισε το έμπολα, τη Φουκουσίμα ή τα χημικά όπλα στη Συρία ή στη Λιβύη οδήγησε πολλούς ειδήμονες στο εξής κανένα καν, κράτος ούτε στο δυτικό ούτε στον αναπτυσσόμενο κόσμο είναι εντελώς προετοιμασμένο σήμερα να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τέτοιες απειλές. Και όντως, εάν κοιτάξουμε τις κρίσεις αυτές, μπορούμε να πάρουμε τέσσερα μαθήματα. Πρώτον, οι πληθυσμοί συχνά είναι κακώς ενημερωμένοι για τις απειλές από χημικές, βιολογικές και ραδιοπυρηνικές ύλες. Δεύτερον, δεν υπάρχει επαρκής προστασία των υποδομών και ειδικότερα από βιολογικές και χημικές απειλές. Τρίτον, η επιβολή του νόμου και οι σχετικές αρχές πολλές φορές δεν έχουν την κατάλληλη εκπαίδευση για να ανταποκριθούν στα καθήκοντά τους σε εποχές κρίσης. Και τρίτον, και πιο σημαντικό, είναι πως η πολιτική ευαισθητοποίηση θα μπορούσε να βελτιωθεί. Αυτά τα τέσσερα διδάγματα δεν πρέπει να μας εκπλήσουν. Τέτοια συμπεράσματα σχετικά με τις χημικές, βιολογικές και ραδιοπυρηνικές απειλές γίνονται συχνά. Τρίτον, η απάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης η αναγνώριση των συνεπειών μιας ανεπαρκούς προετοιμασίας για τέτοια περιστατικά οδήγησε την Ευρωπαϊκή Ένωση στο να αποφασίσει να αναλάβει ευθύνη σε δύο επίπεδα και να δράσει σε δύο επίπεδα. Πρώτον, στο στρατηγικό επίπεδο. χημικέ βιολογικέ και ραδιοπυρηνικέ απειλέ αποτελούν τμήμα τη παγκοσμία στρατηγική τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προετοιμάζει επί του παρόντο μια ανακοίνωση για τι χημικέ βιολογικέ και ραδιοπυρηνικέ απειλέ, που θα ολοκληρωθεί το τέλο του 2016 και θα αναφέρει περισσότερα σχετικά. Την ανακοίνωση αυτή θα ακολουθήσουν σχέδια δράση για την πρόληψη, την ανείχνευση και την αποκρίση. Και στο στρατηγικό επίπεδο υπάρχει η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Βερσοβία τον Ιούλιο του 2016 που αποκαλείται στην ως δήλωση ανθεκτικότητας και αναφέρεται ρητό σε τέτοιες απειλές. Αυτά όσον αφορά το στρατηγικό τμήμα της απόκρισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε επιχειρησιακό επίπεδο. Η ευρωπαϊκή επίπτωση η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ξοδέψει 500 εκατομμύρια ευρώ μεταξύ 2010 έως 2020 για να αναπτύξει εντός και εκτός Ευρώπης ασφάλεια σχετικά με χημικές, βιολογικές και ραδιοπυρηνικές απειλές. Μέσω των κέντρων αριστείας γίνεται η υλοποίηση σε 55 χώρες και 8 περιφέρει, ο περιοχές, τεσσάρων εκ των οποίων στην εγγύ μας περιοχή έχουν ήδη υιοθετηθεί σχέδια δράσης. Θα, θα προσπαθήσουμε να συνεχίσουμε να προσεγγίζουμε χώρες όπως το Ιράν, το Πακιστάν, την Αίγυπτο και το Ισραήλ, καθώς έχουν δείξει ενδιαφέρον για την πρωτοβουλία. Μόνο η διεθνή συνεργασία μπορεί να επιφέρει λύσεις για ένα ζήτημα πολιτικής προστασίας, το οποίο δεν γνωρίζει σύνορα και απαιτεί διεθνή αλληλεγγύη. Μιλώντας για διεθνείς εταιρικέ σχέσεις, επιτρέψτε μου να τελειώσω με μία παρατήρηση. Οι συμπράξεις ιδιωτικού και δημόσιου τομέα θα αποτελούν προαπαιτούμενο στο μέλλον για τον καλό συντονισμό μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα ιδίω σε τομείς όπως είναι οι χημικές, βιολογικές και ραδιοπυρηνικές απειλές. Η χημική βιομηχανία, η φαρμακευτική, επίσης πρέπει να εγκίνουν το συντονισμό τους με τα κέντρα αριστείας και το δίκτυο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η γενική προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο ζήτημα αυτό έχει γίνει αντιληπτή και επικροτήθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, από το ΝΑΤΟ, του G7, G7 και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχει επιβεβαιωθεί πως η προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι υγιής και έχει έναν καλό αντίκτυπο για την ενίσχυση της άμυνάς μας. Μόλις επέστρεψα από τη Νέα Υόρκη, όπου σχεδιάζεται για του χρόνου ένα ψήφισμα των Ηνωμένων Εθνών για τα χημικά, βιολογικά και ραδιοπυρηνικά όπλα, όχι μόνο για την πολιτική ευαισθητοποίηση σχετικά με το ζήτημα αυτό, αλλά επίσης για να χρησιμοποιηθεί η μέθοδος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να επεκταθεί σε άλλους τομείς όπως είναι οι απειλές από τον κυβερνοχώρο. Το ζητούμενο τώρα είναι να εντείνουμε περισσότερο και συντονισμό μας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να δημιουργηθούν συνέργειες μεταξύ εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής μας για χημικά, βιολογικά και ραδιοπυρηνικά όπλα, έτσι ώστε να δημιουργηθεί μια ισχυρότερη ανθεκτικότητα και να αντιμετωπιστεί μια απειλή η οποία δεν πρόκειται να φύγει. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε ο κύριος Μπέντο Σίλβα από την ε, Γενική Διευθύνση Home. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ και όλους σας για την ευγενική πρόσκληση και τον κύριο Ντιπρέ για την διεξοδική του παρέμβαση, με την οποία, στην οποία προσυπογράφω πλήρως. Από την Γενική Διεύθυνση Home, σαφώς επικεντρωνόμαστε κυρίως στις ε, σχεδιασμένες επιθετικές δράσεις με τέτοιου είδου όπλα, ιδίως τρομοκρατία, και στη Γενική και στην Επιτροπή γενικότερα έχουμε μια ε, αντιμετώπιση για τους κινδύνους συγκεκριμένη και για την ε, περίπτωση των χημικών, βιολογικών και πυρηνικών όπλων, ώστε να έχουμε την, ε, έτοιμη την απόκρισή μας και την πρόβλεψη σε αυτές τις περιπτώσεις, όπως και όλα αυτά που ανέφερε ο κύριος Ντιπρέ. Ε, σε ό,τι αφορά τώρα τους κινδύνους. Συμμεριζόμαστε τις ανησυχίες σας. Ιδίως για τους κινδύνους που έχουν να κάνουν με τρομοκρατικές απειλές. Παρακολουθούμε πολύ στενά και κάνουμε στην Ίνσεν και στην ΣΕΑΚ ε, τις, ε, παρακολουθούμε τις δικές τους αξιολογήσεις καθώς και τι κάνουν οι υπόλοιποι διεθνή μας εταιρείοι όπως ε, το ΝΑΤΟ, οι Ηνωμένες Πολιτείες και άλλοι τα υπόλοιπα κράτη-μέλη. Υπάρχει μια σύγκληση διαρκώς προκύπτουν λεπτομέρειες καθώς εξερευνούμε ε, αχαρτογράφητες περιοχές και παρακολουθούμε πολύ προσεκτικά τη δράση τρομοκρατικών ομάδων για να καταλάβουμε τι κίνδυνος υπάρχει για τη χρήση τέτοιων όπλων. Με ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον βέβαια, με το βλέμμα στραμμένο κυρίως στα χημικά, αλλά και στις δυνατότητες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει αρμοδιότητα στην αξιολόγηση του κινδύνου, όμως ακούσαμε μεγάλη προσοχή όσο υπόθηκαν και έχουμε παρακολουθήσει τις ενδείξεις ότι το ISIS έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει κάποια χημικά όπλα όπως ε, με έχει καταγγείλει ήδη το ΝΑΤΟ. Βεβαίως η, ποιότητα αυτών ε, είναι ακόμα που κάτι δεν μπορούμε να αξιολογήσουμε από ιστορικής σκοπιάς τώρα, οι δικές μας πολιτικές για τα χημικά, βιολογικά και πυρηνικά όπλα χαρακτηρίζονται από κάποιες ε, περιόδους. Η πρώτη ξεκίνησε το 2005, μετά τις επιθέσεις στη Μαδρίτη και το Λονδίνο. Εκεί προβλέψαμε, ήδη από νωρίς, κάποιες προβλέψεις για τα όπλα ε, ήδη από το 2005. Με ομάδες εργασίας να ασχολούνται με τον καθένα τομέα ξεχωριστά. Χημικά, βιολογικά, ραδιενεργά, πυρηνικά. Ως προεδρεύων στο Συμβούλιο εκείνο το διάστημα, το 2007, είχα τη χαρά, βάσει της δουλειάς που είχε γίνει προηγουμένως από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να ασχοληθώ με τα θέματα αυτά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν δεν θα έλεγα ότι καμαρώνει ακριβώ, αλλά έχει μια αυτοπεποίθηση γιατί ήδη από τα πρώτα στάδια τη διαδικασία, με τη συμμετοχή του Ευρωκοινοβουλίου, καθώ συζητήσει άρχισαν εδώ πριν από δεκαετία, ε, έχουμε κάποια πείρα στα θέματα αυτά. Στην πρώτη λοιπόν περίοδο έγιναν κάποιε προσπάθειε να είμαστε ε, διεξοδικοί στην ε, κάλυψη των θεμάτων. Δηλαδή τα πρώτα έγγραφα που καταρτίστηκαν προσπάθησαν να επισκοπήσουν όλα τα επιστημονικά στοιχεία που υπήρχαν, ε, στοιχεία από τις εταιρείε, από, τους πολιτικές, από τις υπηρεσίες ε, πολιτικής, από τις ε, διοκτικές αρχές. Δεν θα μπορούσε κανείς να μας καταγορήσει για έλλειψη φαντασίας. Και η βασική μας μέρημνα ήταν η διεξοδικότητα και το κατά πόσο ήταν πλήρη τα στοιχεία. Αυτό οδήγησε στην κατάρτιση προγραμμάτων δράσης Και το πρώτο περιλάμβανε 124 προτεραιότητες. Μάλλον, όταν έχει κάνει 124 προτεραιότητες, καταλήγει να μην έχει καμία και θα μπορούσε να κατηγορηθεί γι' αυτό, αλλά θέλαμε να είμαστε διεξοδικοί, όπως είπα. Και αυτό ήταν μια επιλογή που έγινε. Ε, τα κράτη-μέλη το επέλεξαν αυτό. Δεν θέλαμε να χάσουμε τίποτε από ε, τις ε, διάφορες περιπτώσεις που μπορεί να προέκυπταν. Το πρόγραμμα αυτό εφαρμόστηκε σχεδόν πλήρω, με 66 οριζόντιες δράσεις οι οποίες επιτυχώς ολοκληρώθηκαν. Έχουμε κάνει πράγματα όπως την ε, συμπίληση λεξικού για τα χημικά, βιολογικά, ραδιενεργά, πυρηνικά όπλα που έχει μεταφραστεί σε όλες τις γλώσσες, με ε, δυνατότητες να κατεβάσει κανείς άρθραξ από το ίντερνετ, με τους επαγγελματίες να μπορούν να μιλήσουν μεταξύ τους ε, σε ένα φόρουμ, με τη δεύτερη έκθεση για την εφαρμογή του προγραμματος δράσης ε, για τα όπλα CBRN, το οποίο θα, μετα... θα αποσταλεί στα θεσμικά όργανα, μάλλον ταυτόχρονα με την ανακοίνωση που αναφέρε και ο συνάδελφος. Και έτσι θα μπορέσετε να δείτε συνολικά την κατάσταση και το πώς προχωρούν τα μέτρα που έχουν, επιβληθεί, που έχουν αναλυφθεί. Πάντως, στην ουσία έχουμε ξεκινήσει την ε, εφαρμογή. Η προηγούμενη περίοδος ξεκίνησε περίπου πριν δύο χρόνια και είχε να κάνει με τον ανανεωμένο ενδιαφέρον των Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων, του Κοινοβουλίου συμπεριλαμβανομένου, στα ε, όπλα CBRN και έχει να κάνει με την χρήση χημικών όπλων στη Συρία, για να μην κρύβομαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Η χρήση χημικών στη Συρία έφερε στην πολιτική προσοχή, στο πολιτικό προσκήνιο, τις πιθανότητες τρομοκρατικών επιθέσεων και το συσχετισμό μεταξύ τρομοκρατών, ε, όπλων και της περίπτωσης οι τρομοκράτες να αρχίσουν να αναγνωρίζουν και να χρησιμοποιούν χημικά. Έκτοτε, εκδηλώθηκε ενδιαφέρον στο Συμβούλιο, ήδη από τα συμπεράσματα του Συμβουλίου του 2012, τα οποία πρόλαβαν την χρήση των χημικών. Όμως από το 2014 ως σήμερα επικεντρωθήκαμε πολύ στο αναθερμασμένο ενδιαφέρον των κρατών μελών και του Συμβουλίου για να αναλυφθεί δράση. Έτσι κινηθήκαμε σε πέντε κατευθύνσεις. Ζητήσαμε από τους συναδρέφους της ΑΕΔ και των υπόλοιπων ερευνητικών κέντρων και το κέντρο στρατηγικών μελετών να ασχοληθούν με το έβρος και το βάθος των επιθέσεων ή τις ενδεχόμενες απειλές. Η τι ενδεχομενες απειλες πτυχή ήταν να αναλύσουμε τα γενεσιουργά αίτια των ε, του λαθρεμπορίου ενδεχομένως χημικών με τις θαλάσσιες και χερσαίες οδούς ε, της Μεσογείου και των Βαλκανίων να είναι οι πρώτοι διάδρομοι, οι πρώτες ε, διαδρομές που μας απασχόλησαν. Δηλαδή συνειδητοποίησαμε ότι πρέπει να προσέχουμε, να, έχουμε, να είμαστε σε επιφυλακή στα σύνορα στις περιοχές διέλευσης ε, για την όλη κυκλοφορία των χημικών. Έπειτα θελήσαμε να αναθερμάνουμε τις δραστηριότητες διάφορων ομάδων εργασίας εσωτερικός. Εξωτερικός οι συνεργάτες μας επίσης ήταν ιδιαίτερα δραστήριοι σε διάφορους τομείς αριστείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πάντως, εντός, ε, κοιτάξαμε να αναθερμάνουμε τις διάφορες ομάδες εργασίας και την όλη μας δουλειά για αυτά τα θέματα ώστε να αρχίσει πάλι να παίρνει μπρο το μηχάνημα και να κινηθούμε γρήγορα εφόσον χρειαστεί. Τέταρτον, μαζί με του συναδέλφου τη Γενική Διεύθυνση και πολλά κράτη-μέλη, οργανώσαμε μια μεγάλη προσπάθεια το 2014 με 600 συμμετέχοντες, 7 κράτη-μέλη και η πρώτη άσκηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο ήταν αυτή που έφερε κοντά τι ειδικέ δυνάμει. στους υπευθύνους προστασίας των πολιτών. Απολύμανση, ιατρικές ε, καταστάσεις, ιατρικά προγράμματα μάλλον, ελεύθεροι σκοπευτές. Σε ένα πολύ πολύπλοκο σενάριο, με ομήρους, με αναπαράσταση οι εμπειρογνώμονες ε, είδαν κατά πόσο μπορούν εγκαίρως να εντοπίσουν τους ουσίες, να προλάβουν τη μετάδοση, ε, με την παρεμβολή των ε, πρακτόρων, ασφάλειας. Όλα αυτά ήταν ιδιαίτερα περίπλοκα, αλλά καταφέραμε να τους συνδυάσουμε και με τρόπο χειροπιαστό να προσελκύσουμε την προσοχή των πολιτικών ηθινόντων. ώστε όλα αυτά να ειδωθούν από κοινού θέλαμε να δείξουμε ότι έχουμε κάνει πολλά, ότι έχουμε τα εργαλεία εν γέννη για να ανταποκριθούμε σε τέτοιες καταστάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ότι δεν βρισκόμαστε σε φάση άγνοιας, ούτε ε, φλούμε. Δεν έχουμε και επειδή πολύ νωρί ε, ε, έγιναν πολλά ήδη. Έχουν ακόμα πολλά να γίνουν. Το πέμπτο λοιπόν στοιχείο ήταν μια προσπάθεια να εξευρεθούν αποδεκτικά στοιχεία και να δούμε πού έχουμε φτάσει, πώς έχουμε προχωρήσει και τι πρέπει να γίνει τώρα κατεπηγόντως προτού ξανασχεδιάσουμε και, ξανα, ε, και ανακατευθύνουμε την πολιτική μας και τους στόχους της. Είδαμε σε ποιου τομεί δεν υπάρχει στρατηγική πρόοδος και που πρέπει να κινηθούμε. Ε, μεταξύ των απειλών των κινδύνων και άλλων. Την ανακοίνωση την έχετε λάβει και την έχετε μελετήσει, υποθέτω, οπότε ξέρετε γιατί μιλάω. Προβλέψαμε λοιπόν αμέσως μια σειρά από δράσεις και είπαμε ότι πρέπει να γίνει διεξοδική ανάλυση του τι συμβαίνει στην πράξη. Γι' αυτό υποβάλαμε και ένα έγγραφο για την κατάσταση που προβλέπεται να επικρατήσει από στατηγική σκοπιά στο ερχόμενο διάστημα. Όπως θα ξέρετε, υπήρξαν πρόσφατες εξέλιξεις που επηρεάζουν την προετοιμασία αυτής της ανακοίνωσης. Θα προσπαθήσω να ολοκληρώσω σε ένα-δυο λεπτά. Εξορισμού Μιλάμε για μια απίστευτα περίπλοκη περιοχή μελέτης. εμπλέκονται ένα σωρό γενικέ διευθύνσει, το Κοινό Κέντρο Ερευνών, εμεί οι ίδιοι, το Ευρωκοινοβούλιο και όχι μόνο ω στο ρόλο του νομοθέτη, η δουλειά τη Γραμματεία του Κοινοβουλίου, η έκθεση που δημοσιεύτηκε το Γενάρη και επικαιροποιήθηκε το Μάιο, έχουμε ε, συμβάλει έχω συναντηθεί με βουλευτές, έχω συζητήσει μαζί τους Το κοινοβούλιο λοιπόν δεν ήταν απλώς αποδέκτης, ήταν και ε, δρόν πρόσωπο στην όλη διαδικασία. Πρέπει λοιπόν να ε, αξιοποιήσουμε τις ιδέες που προσφέρονται σε όλο αυτό το στοχασμό μας και με τον νέο επίτροπο, τον Τζούλιαν Κίνγκ για την Ένωση της Ασφάλειας και με την ομάδα δράσης όπου συνδυάζονται οι τρεις γενικές διευθύνσεις και η ΕΕΔ. Δεν θέλουμε να μας λείψει τίποτα στην όλη προσπάθεια από τα απαραίτητα στοιχεία για να καταλήξουμε στο αποτέλεσμα μας ένα τόσο περίπλοκο τομέα. Κοιτάζουμε λοιπόν μπροστά στο μέλλον και θέλουμε να είμαστε βέβαιοι ότι θα εκμεταλλευτούμε όλα τα πλεονεκτήματα που έχουμε και ότι θα αξιοποιήσουμε όλη την πολιτική βούληση όλων των ε, ενδιαφερομένων θεσμών. Η ανακοίνωση που θα δημοσιεύαμε το Δεκέμβρη, ίσως να προκύψει το Γενάρη το Φλεβάρι, δεν θέλει ότι από τώρα δεν θα είναι έτοιμη το Δεκέμβρη, λέω απλώς ότι έχουμε νέους πολιτικούς ηθήνοντες και έχει δοθεί ε, πλήρης προσοχή σε μια σειρά από προοπτικές που ως τώρα ήταν πολύ δύσκολο να τις συνδυάσουμε. Αλλά τώρα αυτό έχει καταστεί πλέον εφικτό. Γι' αυτό είμαι βέβαιος ότι σε λίγους μήνες θα μπορούμε να επανέλθουμε στο Ευρωκοινοβούλιο, σε αυτή την Επιτροπή και αλλού, και στην Επιτροπή ΛΥΜΠ μάλλον και να παρουσιάσουμε τις ιδέες της ανακοίνωσης. Και πάλι σας ευχαριστώ πολύ κυρία Φωτίγκα για την ευγενική σας πρόσκληση. Εμείς σας ευχαριστούμε. Ναι, πράγματι δεν ε, υπάρχουν και πολλά χρονικά περιθώρια και είναι καλό να μας βοηθήσετε κι εσείς. Έχουμε να δούμε την ε, τεκμηρίωση και τα επόμενα έγγραφα που έρχονται. Θα πρέπει να μελετήσουμε και αυτά. Uh, I think there are Υπάρχουν νομίζω κάποιοι βουλευτέ. Μάλιστα, ο κ. Γκάλερ. Ευχαριστώ. Θέλω να σας ευχαριστήσω για αυτή την παρουσίαση των διαδικασιών. Είπατε, είπατε πολύ σωστά ότι και εμείς στο Κοινοβούλιο από έχουμε ασχοληθεί. Έχω μπροστά μου την έκθεση Αναγκόμης από το Δεκέμβριο του 10 με έναν κατάλογο διεκδικήσεων που είχαμε, κάποιων ετοιμάτων που είχαμε διατυπώσει. Να σας πω λίγα. Ποιοτικά πρότυπα, πρότυπα ασφαλείας, νέο σύστημα και δίκτυο εργαστηρίων για την πιστοποίηση εξοπλισμού ασφαλείας και τεχνολογιών, CBRN ή κάτι άλλο που ζητάμε, τι είναι για να το βρω. Ανταλλαγή, χρήση, βέλτιση των πρακτικών, γνώσεων, τεχνογνωσίας από το τομέα της στρατιωτικής και μη στρατιωτικής ε, χρήσης κτλ. κτλ. Ασφαλιστικές δικλείδες, μέτρα ασφαλείας, με τις ε, βάσεις δεδομένων και τα ευαίσθητα δεδομένα. Θα μπορούσα να συνεχίσω να μιλάω για ώρες αλλά αυτά τα ζητούσαμε το 10. Πολλά έχουν υλοποιηθεί έκτοτε, οπότε το ερώτημά μου είναι... Επειδή αναφερθήκατε εδώ στα θεσμικά όργανα που συνεργάζονται, τι ωραία, τι καλά. Τα κράτη-μέλη όμως είστε ικανοποιημένοι από τη δική τους ε, συνεργασία και συμμετοχή στις προσπάθειες που βλέπετε περιθώρια βελτίωσης στο κοινοβούλιο, ξέρετε, μπορείτε να κατονομάσετε τα κρατημέλη. Ξέρω ότι δεν σας αρέσει να το κάνετε, αλλά κάποιες φορές καλό είναι να ονομάζουμε για να ονειδήσουμε. Ποια επικοινωνία υπάρχει σε επίπεδο, μεταξύ Ευρωπαϊκού και Εθνικού επίπεδου. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ κύριο Καν. Ναι, θέλω να ευχαριστήσω και εγώ για τις πληροφορίες. Δεν ξέρω αν κατάλαβα καλά όμως. Για το ίσες και το ΝΤΑΕΣ που είναι το ίδιο πράγμα. Είπατε ε, κάτι για χημικά όπλα. Δηλαδή τι θα πει αυτό. Μπορούν να τα παρασκευάσουν ή έχουν αποθέματα από το Ιράκ και τη Συρία. Αυτό το ένα και το δεύτερο που σχετίζεται με το πρώτο. Είδαμε ότι Πιέζεται από παντού τον ΤΑΕΣ. Σε σχέση με τα χημικά όπλα, τι σχέση βλέπετε. I'm not sure whether... Ο κύριος ε, Σαφοζέ θέλει το λόγο. Όχι, άρχισα πολύ, συγγνώμη. Μάλιστα, λέει ο πρόεδρος. Να κάνω κι εγώ μια ερώτηση. μια δήλωση μεταξύ ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν κάποια πλάνα. Μπορείτε να μας πείτε τίποτε. Υπάρχουν άμεσα σχέδια. Θα αλλάξει αυτή η δήλωση το τρόπο συνεργασίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ. Θα τολμούσατε να πείτε έτσι μια πρόσθετη ερώτηση σε σχέση με το που βρισκόμασταν πριν 10 χρόνια και το που είμαστε σήμερα. Θα τολμούσατε να πείτε ότι είναι πιο ασφαλή ήδη οι πολίτε μα με τα μέτρα που έχουν ληφθεί. Κύριοι, έχετε το λόγο, λέει πρόεδρο. Ίσως με την ίδια σειρά. Right. Συμμετοχή των κρατών μελών. Εγώ μπορώ να μιλήσω μόνο για την εξωτερική πτυχή. Το 80% περίπου της χρηματοδότησης για τα κέντρα επιστρέφει στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί για δική τους εμπειρογνωμοσύνη, εμπειρία και τεχνογνωσία πρόκειται. Έχουμε δημιουργήσει κοινοπραξίες από κράτη-μέλη, ΜΚΟ, αν έχουν την εμπειρία, γιατί είναι ένα πολύ το τομέας αυτό και επίσης έχουμε προσπαθήσει να διευρύνουμε το πεδίο της συμμετοχής των κρατών μελών. Όταν ξεκίνησε το 12 η πρωτοβουλία αυτή, τρία πέντε κράτη-μέλη είχαν την δυνατότητα δεν μπορώ να σας πω τα ονόματα βέβαια, αλλά έρχονται και άλλα τώρα. Γιατί έχουν ε, μάθει για τις διαδικασίες ε, και έχουν βελτιώσει και τις δυνατότητες αντίδρασης ε, για τα CBRN και τη βοήθεια από τρίτες χώρες για δήλωση ΝΑΤΟ Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πολύ νωρίς Έχουμε ξεκινήσει τις διαπραγματεύσεις, αλλά ε, και εντός η και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αρχίζουμε λοιπόν και συζητάμε ήδη τι μπορούμε να βελτιώσουμε, τις λεπτομέρειες. Δεν μπορώ να σας δώσω όμως τώρα κάποια πληροφορία, απλά αρκεί να πω ότι υπάρχουν κάποιες επαφές υπαλλήλων από το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είχαμε ε, στο Βιτσκόφ επαφή και από κάποια για το CBRN και θα δούμε πώς μπορούμε να ενισχύσουμε τη σχέση. Ο επόμενος. Ευχαριστώ. Με τη σειρά να απαντήσω στα ερωτήματα. Η έκθεση της Άννα πόσο ε, μέρος της έχει ήδη υλοποιηθεί. Πρώτον, όταν ανέφερα Πολλέ δραστηριότητε ότι γίνονται εδώ στο Κοινοβούλιο, συναντήσει με ευρωβουλευτέ που ενδιαφέρει το θέμα. Η Αναγκόμες είναι και συμπατριώτησά μου και είναι μία από ε, αυτούς ή αυτές που δείχνει ε, έντονο ενδιαφέρον και με πολύ χαρά συνεχίζουμε τις συζητήσεις μαζί της, αλλά και μάλιστα τη Μόνικα Χολμάγερ και πολλούς άλλους. Τα συγκεκριμένα παραδείγματα που δώσατε τώρα ό,τι αφορά την πιστοποίηση, ό,τι αφορά συνεργασία στρατιωτικού με στρατιωτικού τομέα. Θετική είναι η απάντηση που μπορώ να σα δώσω, καταφατική. Ευτυχώ δεν ρωτήσατε άλλα, ήμουν τυχερό. Αλλά για αυτά τα δύο κάναμε πράγματα. Είναι οριζόντιο το θέμα. Δηλαδή, έχουμε τη γνώση των χρηστών της τεχνολογίας, τον κύκλο της ε, γνώσης. Πώς όλα αυτά τα βάζουμε μαζί. Υπήρχαν τα SRAB, SRIF, 600 εμπειρογνώμονες ε, για να βρουν στρατηγικούς τρόπους ε, να συνδυάσουν ανάγκες και δυνατότητες Εμείς είχαμε επαφές και μιλήσαμε με κάποιους που υποστηρίζουν αυτές τις ε, προσεγγίσεις, ακολουθήσαμε όμως μια προσέγγιση από κάτω προς τα πάνω. Αυτές οι ομάδες που σας είπα, για τα βιολογικά χημικά λοιπά, εμπειρογνώμους των μελών, με αυτού, λοιπόν προσπαθήσαμε να ξεκινήσουμε δραστηριότητες με συμμετοχή και άλλων εμπειρογνωμόνων από άλλους κλάδους από αυτούς που είχαν να κάνουν πιο πολύ με την ασφάλεια μέχρι τους που είχαν πιο πολύ με την τεχνολογία για να ε, συγκεντρώσουμε καλές πρακτικές ε, να δούμε τις ε, επιδόσεις τις πραγματικές και από εκεί να βρούμε μια βάση για πιθανές δραστηριότητες πιστοποίησης, τυποποίησης. Δεν ξέρω, ίσως πίσω οι συνάδελφοι να ξέρουν. Νομίζω είναι 7 δραστηριότητες τυποποίησης στον τομέα της εντοπισμού και προστασίας που άμεσα προέρχονται από την κοινή δουλειά των κρατών μελών και των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Διότι εντοπίστηκαν με τον τρόπο αυτό καλέ πρακτικέ. και έτσι οι φορεί πιστοποίηση έχουν στοιχεία για να προχωρήσουν στι πιστοποίησει. για τι επιδόσει των εργαλείων και για την τυποποίηση και και για την πιστοποίηση. Η συνεργασία μα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνα. συνεχίζεται και καλύπτει διάφορου τομεί. ΣΥΑΚ. Φυσικά χρειάζεται στρατιωτική εμπειρία για την αξιολόγηση κινδύνων και απειλών. Βέβαια υπάρχουν περιορισμοί. Προφανώς υπήρχαν και με τη συνθήκη τη Λισαβόνα. το στρατιωτικό και με στρατιωτικό σκέλος πρέπει να ε, συνεργαστούν περισσότερο. Όμως οι συνάδελφοι που ασχολούνται με τα συμπεράσματα και τα εκρηκτικά έχουν συχνά επαφέ με διαφόρου ειδικού από διάφορου τομεί. και φραγμοί που υπήρχαν σε, στη σχέση στρατιωτικού με στρατιωτικού σκέλους ε, υπερπηδούνται σιγά σιγά. Να σα δώσω ένα παράδειγμα. Ή μάλλον να αφήσω τελευταίο το τελευταίο ερώτημα που είναι και το πιο δύσκολο. Αν είναι πιο ασφαλεί πολίτε μας. Να πέρασω τον κύριο Καν. Νταέ, τι δυνατότητε έχει. Εμείς Είμαστε αποδείκτε και όχι αυτοί που παράγουμε τι αξιολογήσει απειλών και κινδυνών, αλλά δεν μπορώ να κάνω κρίση και αξιολόγηση. Αλλά όλη η δουλειά που γίνεται για την αξιολόγηση κινδύνων από CBRN, όπλα, βασίζεται στο ότι πιστεύουμε οι πληροφορίες που λαμβάνουμε από διάφορες πηγές, ότι ο Ντάι μπορεί να χρησιμοποιήσει αφού τα παραγάγει ε, χημικά όπλα, ε, είναι πληροφορίες για τις οποίες δεν μπορούμε να, ξέρουμε, δεν γνωρίζουμε τις πηγές όταν είναι ασφαλείς, αλλά το λαμβάνουμε υπόψη μας. Για ε, διάφορα αέρια ε, που μπορεί να παραγάγουν και αν μπορούν αυτά τα αέρια να τα χρησιμοποιήσουν ως όπλα. Διεθνή συνεργασία. Για να συμπληρώσω αυτό που και ο κύριος Διπρέ. Πολλοί συνεργάζονται ο συνάδελφος που κάθεται πίσω και παίρνει σημειώσεις ήταν στις ΗΠΑ την προηγούμενη εβδομάδα μαζί με το αφεντικό του τον προϊστάμενο το τμήματος για τα όπλα CBRN και συναντήθηκαν με διάφορους εμπειρογνώμονε από πολλούς φορείς. Στόχο ήταν η προετοιμασία του follow-up τη συμφωνία τη Υπουργική ε, συνάντησης ε, για τα θέματα CBRN και το τι θα γίνει θα το γνωρίζουμε περισσότερο στους επόμενους μήνες. Είχαμε ενισχυμένους πολιτικούς διαλόγους και με άλλες χώρες όπου το, τα όπλα CBRN συζητούνται ρητός, άρα εξωτερική διάσταση της εσωτερικής ασφάλειας εντάσσεται στις προσπάθειες και είναι συμπληρωματική ως προς ε, τις ε, ε, χρηματοδοτικές προσπάθειες, μία, DEFCO, και άλλο και η πατή εκπρόσωπος Μουγκερίνη και εμείς έχουμε επαφές με τους ε, ομολόγους μας από τρίτες χώρες που έχουν εμπειρία για τα όπλα συμπιάρια. Αν το επιτρέπει βέβαια το πολιτικό πλαίσιο, που το επιτρέπει βέβαια, σε ό,τι αφορά τη ΣΥΠΑ τουλάχιστον. Όχι όμως με όλες τις χώρες του κόσμου. Δεν θα μπορούσαμε αυτές να έχουμε, με όλες αυτές να έχουμε τόσο εκτεταμένη συνεργασία. Το τελευταίο στοιχείο της ερώτησης του κυρίου Γκάλερ τώρα, για να απαντήσω, δεν ξέρω. Δεν είμαι βέβαιος ότι μπορώ να σας απαντήσω. Τι μπορώ να πω με τα βεβαιότητος. Ότι οι κίνδυνοι, ιδίως για βιολογικά, για φιλικές απειλές, Εμείς πήραμε την πρωτοβουλία και πριν από 10 χρόνια μάλιστα, μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δηλώσαμε ότι βλέπαμε ότι θα υπάρχει δυνητικός κλιμάκωση ε, των βιολογικών απειλών μέσα σε πέντε χρόνια που μπορεί να είναι ανεξέλιξη ως εξέλιξη. μειωνόταν η τιμή, ε, αυξάνονταν οι φοιτητέ ε, σε μεταπτυχιακά, δακτορικά. Τότε είχαμε πάνω 5.000 εταιρείε που μπορούσαν να χειριστούν τέτοιε ουσίε και ούτω καθεξής. Έκτοτε, κάποια στοιχεία που από πολιτική και επιστημονική πλευράς φαίνονταν ε, φανταστικά, ε, επιστημονική φαντασία, τα λεγόμενα bio garage, ότι δηλαδή θα μπορούσε πάρα πολύ εύκολο οποιοδήποτε ε, πολίτης να παίξει με πάρα πολύ ακριβή και ακριβό εξοπλισμό Τελικά υπήρξε αντίδραση υγιής από, τους, ε, από τα κράτη-μέλη. Ενδιαφέρονται και οι απλοί πολίτες για την επιστήμη και για τις επιστημονικές τεχνολογικές δυνατότητες πήραμε στο μέλλον. Με όλες τις ισχυρές τεχνολογίες όμως έρχεται και η απειλή, ο κίνδυνος μαζί. Για να είμαι απόλυτη ειλικρινής λοιπόν, μπορώ να σας πω ότι αν δεν είχαμε δράσει τότε, οι δυνητικοί κίνδυνοι θα μπορούσαν να είχαν επιδεινωθεί ανεξέλεγκτα σε εκείνη την περίοδο. Αλλά με έγκαιρες προληπτικές δράσεις και με την κινητοποίηση των κρατών μελών που δεν είχαν ακόμη αντιληφθεί τον κίνδυνο, συγκρατήσαμε τις εξελίξεις. Άρα οι απειλές είναι πολύ πιο μέτριοπαθείς σε σχέση με το τι θα είχε γίνει αν δεν είχαμε δράσει εγκαίρως. Για να απαντήσω όμως ε, με πλήρη τρόπο, δεν μπορώ. Είμαστε πολύ καλύτερα προετοιμασμένοι, έχουν αυξηθεί όμως οι κίνδυνοι και απειλές. Το να πούμε ότι είναι πολύ πιο ασφαλείς οι πολίτες μας από ότι θα ήταν αν η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ήταν εδώ, 100% ναι είναι απάντηση. Εγώ έχω γράψει έγγραφα που σας το λέω. Έχω προτείνει πολιτικές και στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή. Άρα μπορώ να την υποστηρίξω πλήρω αυτή τη δήλωση. Ότι δεν θα ήταν ε, ασφαλής πολίτε αν δεν υπήρχε Ευρωπαϊκή Όμω οι εξελίξει στη Συρία, στο Ιράκ, η πρόσβαση ε, στο Πανεπιστήμιο τη Μοσούλη, στο Ζαχάροφ, σε έναν άνθρωπο που δεν ζει, δεν συνεργάστηκε για την προσπάθεια ε, δημιουργίας ε, βιολογικών όπλων το Πανεπιστήμιο της Μοσούλης και ο συγκεκριμένος το πλήρωσε από το Πανεπιστήμιο τη ζωή του αυτό που δεν συνεργάστηκε με τον Τάις για τις ε, όχι βιολογικές αλλά ραδιενεργές ουσίες που ήθελε να αποκτήσει τον Τάις και να φτιάξει όπλα. Άρα η πρόσβαση σε ενεργό υλικό, στην επιστήμη, στα εργαστήρια, οι εξελίξεις από πλευράς ΔΑΕΣ, η αλλαγή πίστης ε, από αυτός που έλεγε για τα όπλα αυτά που πέρασε από την Αλκάιντα στο Δαές. δεν ε, θα ήμουν ειλικρινής και δεν θα καθυσίχαζα ε, ειλικρινός πολίτης αν έλεγα ότι είναι πιο ασφαλής. Απλά θα ε, επαναλάβω ότι αν το Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ήταν εδώ να εφιστά την προσοχή σε αυτά τα προβλήματα, οι πολίτες θα ήταν πολύ λιγότερο ασφαλείς από ότι είναι. Νομίζω η πολιτική ευαισθησία έχει αυξηθεί οι πολιτικές γνώσεις το ίδιο και οι τεχνικές διότι και εντό και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, υπάρχει κόσμος που ασχολείται με αυτά. Όπως είπατε όμως, κύριε Μπέντου Σίλβα, και οι απειλές έχουν ε, πολλαπλασιαστεί και το πόσο περίπλοκες είναι, αν συνδυάσει κανείς κλιματικές αλλαγές με εγκληματικές προθέσεις, με την ενεργειακή ασφάλεια, τη βιοτεχνολογία και την ανατεχνολογία. Έχετε ε, μια συνταγή για φυσικές καταστροφές που μπορούν να συνδυαστούν και με εγκληματικές ενέργειες. Αυτό περιπλέκει τα πράγματα. Ευχαριστώ πολύ. Ε, και οι δύο απαντήσεις ήταν πολύ καλός τρόπος να δώσουμε τέρμα σε αυτή τη συζήτηση. Δεν αισθάνομαι ότι θα πρέπει να πιέσουμε περισσότερο και να έχουμε μια πιο μεγάλη, αποκάλυψη στοιχείων σε αυτή τη ε, ε, συζήτηση που μεταδίδεται στο διαδίκτυο. Κάποια στιγμή ίσω σε μια συνάντηση και κλεισμένων των θυρών. Γιατί το θέμα και επίκαιρο είναι και εξαιρετικά ενδιαφέρον. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους δύο εξέχοντες προκειμένους μας που εκπροσωπούν δύο θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα οποία ασχολούνται με την ε, περαιτέρω οργάνωση της Ευρώπης την αντιμετώπιση τέτοιου τους όπλων. Ευχαριστώ τους Ευρωβουλευτές και τους υπόλοιπους συμμετέχοντες στην αίθουσα για την παρουσία τους και τη συμμετοχή τους σε αυτή τη συνεδρία. Αυτά σας ευχαριστώ, κύριοι μου. Σας αποχαιρετώ και θα περάσω αμέσως στο επόμενο σημείο. Well, business? Ε, λοιπόν, διάφορα. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να σας πληροφορήσω ότι η επόμενη συνεδρίασή μας θα γίνει στις 9 Νοεμβρίου. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την ε, μακρά συνεδρία της Επιτροπής ΕΝΤΑ σήμερα. Ήταν φοβερά ενδιαφέρουσα η συζήτηση και θερμές ευχαριστίες και προς τους διερμηνείς για τη δουλειά τους. Ολοκληρώνω τη συνεδρία σας.